Uh, ladies um, Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω όλους να καθίσετε στις θέσεις σας. Ώστε να ξεκινήσουμε την ειδική συνεδρίαση μισής μέρας εδώ να ξεκινήσω ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους σας. Ελπίζω να τα περάσετε καλά στις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές και να επανήλθατε ανανεωμένοι για να εξετάσουμε τα σημαντικά προγράμματα για τα οποία δουλεύει η Επιτροπή μας. Ε, βασικό μας θέμα απόψε είναι το, η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, πολύ σημαντικό θέμα και να σας θυμίσω ότι στις 4 έχουμε ψηφοφορίες για δύο γνωμοδοτήσεις που, που πρέπει να ψηφιστούν σήμερα, ώστε να περάσουν στην αρμόδια επί της επιτροπή. Είναι η έκθεση της κυρίας Μακάρτιν για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας των προϊόντων του μέτρου δομικών κατασκευών. Ε, και ε, για την ε, έκθεση Κρόιτσμαν για τη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Επίσης θα πρέπει να βρούμε και μια συμφωνία για τα εινοδηγία, για τα δομικά προϊόντα. Καθώς επίσης πρώτα θα μιλήσουμε για την έκθεση για τις ε, πολιτικές επιλογές για το συμβατικό δίκαιο στην Ένωση. Έχω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση να σας κάνω σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Δυστυχώς η συγγήτρια δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, αλλά μου ζήτησε να σας διαβιβάσω το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής μας. Βασικά, όλα τα αιτήματα και οι προτάσεις που προτείναμε στον προπολογισμό έγιναν, αποδεκτέ, έγιναν αποδεκτές στην τελική συμφωνία, δηλαδή υποστήριξη για το πιλωτικό πρόγραμμα για το φόρουμ για την ενιαία αγορά, προπαρασκευαστική δράση στον τομέα της πολιτικής ε, του καταναλωτή, η στήριξη στο Σόλβιτ για μια χωριστή γραμμή του προπολογισμού, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, και κάποια άλλα από τα ζητήματα που είχαμε εμείς αναφέρει. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να κάνει η κυρία Σόλτερ Μόζερ, Α, συγγνώμη, η κυρία Ρούλερ που είναι υπεύθυνη για τον προπολογισμό. Ζητώ συγγνώμη, αν και δεν είναι εδώ για να διαπιστώσετε λάθο μου. Ε, λοιπόν, χρειάζεται να φτιάξουμε ένα σωστό χρονοδιάγραμμα ώστε να έχει η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού τη γνωμοδότησή μα για την απαλλαγή του περασμένου χρόνου. Η κυρία Ρούλε μόλι έφτασε και Χάιντι μιλούσα για την απαλλαγή του 2009 για την οποία είσαι εσύ υπεύθυνη. Μα ζήτησε να φτιάξουμε μια γνωμοδότηση που πρέπει να γίνει αυτή την εβδομάδα, να συζητήσουμε την 1η Φεβρουαρίου και να την υιοθετήσουμε στις 28 Φεβρουαρίου. Θέλεις κάτι να μας πεις? Αυτό αφορά την απαλλαγή σου. Συμφωνείς? Εφόσον όλοι συμφωνούμε να ακολουθήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θες κάτι να προσθέσεις? Όχι. Ωραία. Απαλλαγή λοιπόν της κυρίας, μάλλον η έκθεση για την απαλλαγή για το 2009 θα γίνει με αυτό το χρονοδιάγραμμα και για τα άλλα που σας είπα αφορούν τις προτάσεις για το 2010 που θα ε, το, το έχει αναλάβει η κυρία Σόλτερ Μόζερ. Λοιπόν, α ε, αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση για την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να ακούσουμε τον καθηγητή Μάρτιν Σμιτ Κέσελ, που έχει ετοιμάσει ένα ενημερωτικό έγγραφο για μας για τις πτυχές ε, του ψηφιακού περιεχομένου όσον αφορά την οδηγία αυτή για τα δικαιώματα του καταναλωτή Προτείνω λοιπόν να τον καλέσουμε να μας κάνει την ε, εισήγησή του. Ο εισηγητής μας κύριος Σβάμπ είναι εδώ βεβαίως και διάφορες σκιώδεις καλούνται να σχολιάσουν καθώς και η κυρία Γουόλη, που είναι η συγγήτρια για την Επιτροπή την Νομική και δεν ξέρω και ποιο άλλο θα ήθελε να σχολιάσει. Κύριε Σβάμπ, θέλετε να σχολιάσετε εξ αρχή ή θα περιμένετε να ακούσετε την εισήγηση. Θα περιμένετε με την εισήγηση. Με τα χαρά λοιπόν καλωσορίζω τον ε, καθηγητή Σμιτ Κέσελ. Ξέρω πω έχετε κάποιε διαφάνειε που παρουσιάζουν αυτό το ενημερωτικό έγγραφο. Θα το έχετε, ε, είναι διαθέσιμο και θα είναι διαθέσιμο και στο site μας από την Τετάρτη. Με τα χαράς λοιπόν σας δίνω το λόγο να κάνετε την εισήγησή σας και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια των ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω κάποια κατανόηση γιατί έλαβα την εντολή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και σήμερα το πρωί βεβαίως ε, ήταν η προθεσμία και έδωσα τα σχετικά στη γραμματεία Χθε το βράδυ γιατί είχαμε και Χριστούγεννα, έπρεπε να δω και την οικογένεια κτλ. Θα ήθελα βεβαίω να πω πως ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο με απασχολεί εδώ και καιρό και θα ήθελα για λόγους απλότητας να ξεκινήσω με τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην επόμενη διαφάνεια. Τα θέματα δηλαδή, τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Επιτροπή, τα οποία είναι στα αγγλικά για λόγους απλότητας, βεβαίως εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Το πρώτο ερώτημα είναι εάν θα πρέπει το ψηφιακό περιεχόμενο να αντιμετωπιστεί στην οδηγία ή σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς από τον νομοθέτη. Το δεύτερο ερώτημα στοχεύει στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του να αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό περιεχόμενο στην οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών και βεβαίως ε, η πιο εκτεταμένη ερώτηση είναι βεβαίως το πώς ορίζεται το ψηφιακό περιεχόμενο από πλευράς νομοθεσίας και σε ποια κομμάτια της οδηγίας πρέπει να ενταχθεί. Η απάντηση στα δύο πρώτα ερωτήματα, βλέπετε την επόμενη διαφάνεια, είναι πάρα πολύ σύντομη. Κατά την άποψή μου είναι κάτι το αυτονόητο, δηλαδή πως και τα δύο μέσα και η οδηγία δικαιωμάτων του καταναλωτή και το κοινό πλαίσιο αναφοράς ή το κάτι επιλογή αυτό, το προαιρετικό αυτό μέσο μπορούν να ε, ασχοληθούν με το ψηφιακό περιεχόμενο και αυτό όχι μόνο γιατί πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τομείς ε, που απασχολούν τους καταναλωτές και δραστηριοποιούνται οι καταναλωτές διασυνοριακά και άρα στο πλαίσιο της κοινής αγοράς, αλλά γιατί κυρίως ήδη αποτελούν κομμάτι του κοινωνικού κεκτημένου αυτές οι συμβάσεις και θα έπρεπε να κάνουμε βήμα προς τα πίσω εάν τα αφήναμε αυτά απ' έξω. Όσον αφορά βεβαίως το ζήτημα το βασικό από πλευράς του δικαίου είναι οπωσδήποτε το εάν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή το οποίο νομίζω αποτελεί κάτι το θεμελιώδες στο ε, ευρωπαϊκό δίκαιο προσέγγισης του καταναλωτή αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ψηφιακό περιεχόμενο. Πρέπει λοιπόν να το δούμε ρεαλιστικά και να τεθεί για περιπτώσεις κατ' ουσίαν στην οποία ε, έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με την αγορά, δηλαδή κάποιου είδους μετάδοση. Αλλιώς βεβαίως ε, δεν έχουμε και τόσο σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν δύο πτυχές. Υπάρχει ένας ε, τομέας εδώ πέρα στον οποίο ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά σε αγορές εξ αποστάσεως οι καταναλωτές αλλά πρέπει να λάβουμε επίψεις ε, πάρα πολύ σοβαρά πως θα πρέπει να δούμε πως θα... Ε, δεν θα υπάρξει ζήτημα κατάχρησης, δηλαδή να ασκήσει κάποιος το δικαίωμα επαναχώρησης μετά την παράδοση ε, του προϊόντος. Π.χ. αν ε, πάει κανείς στους φοιτητές και δει τι έχουν στον υπολογιστή τους, ή και σε έναν πατέρα που έχει παιδιά και πάνε στο σχολείο νομίζω πως ε, είναι προφανές και θα πρέπει βεβαίως ε, να ξέρουμε πως ε, ίσως εδώ πέρα ο κόσμος δεν έχει πάρα πολύ κατά το που τελειώνουν τα δικά του δικαιώματα και αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε νομικά. Εξαρτάται από το εάν ο επιτιδευματίας ή ο κατασκευαστής ή ο έμπορος ή όπως θέλετε να το πούμε, εάν έχει την δυνατότητα να προστατευθεί από μόνος του τεχνολογικά. Και βεβαίω ε, αυτά είναι μέσα τα οποία προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί κοπηρά τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Υπάρχουν τέτοια μέσα, η δε προσωπική μου εκτίμηση, αλλά αυτή είναι μια εκτίμηση ε, ε, ενό ανθρώπου βεβαίω, ο οποίο δεν είναι πλήρως αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα είναι πω θα μπορούσε να είναι ε, εφικτή μια τέτοια προστασία, αλλά νομίζω πως εδώ πέρα χρειάζεται απλά μια πολιτική απόφαση και θα μπορέσουμε εδώ πέρα να κάνουμε και μια πρόβλεψη, αν θέλετε, προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Το επόμενο θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα και ως επιστήμονα στην όλη αυτή συζήτηση και νομίζω παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο ορισμός. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου. Νομίζω πως όλες οι νομικές τάξεις των κρατών μελών θεωρούν ή τότε το ψηφιακό περιεχόμενο ως υπηρεσία, κάτι το οποίο νομίζω είναι κάτι το ιδιαίτερα άσχημο, δηλαδή από τεχνική σκοπιά της νομοθεσίας δεν είναι πάρα πολύ θετικό, ανεξαρτήτως των πολιτικών ζητημάτων βεβαίω που εγείρονται. Είναι οπωσδήποτε λάθος το να ορίζεται ως ε, υπηρεσία και δημιουργείται εδώ πέρα μια δυνατότητα να υπάρχει και σύγχυση. Και στην πλευρά της ε, νομολογίας. Οπότε Ούτως ή άλλως ε, εμείς δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ στο γερμανικό δίκαιο πως η μετάδοση παραδείγματος χάρη του software μπορεί να αποτελέσει κάποια παροχή υπηρεσίας. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στην επόμενη διαφάνεια πως βλέπετε πως δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το πώς ακριβώς το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί αντικείμενο της ε, σύμβασης, δηλαδή το πώς θα γίνει η αγορά, ε, το πώς θα γίνει η μεταφορά σε μόνιμη βάση ενός ε, ψηφιακού προϊόντος ή αν θα είναι μόνιμη η χρήση. Μετά υπάρχει η προσωρινή χρήση, οπότε να έχουμε κάποιο είδους ενοικίαση αν θέλετε και βέβαιως η μεταφορά με την χρήση ψηφιακών μέσων ε, όπως το streaming, ε, video on demand κτλ. Αυτά πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Δεν το κάνει αυτό μέχρι στιγμής η πρόταση γιατί όλες αυτές ε, οι μορφές όπως σας είπα δυστυχώς έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες και αυτό είναι λάθος και πρέπει νομίζω να είναι σαφές πως ε, πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία επιτρέπει νομίζω κάποιες παρεμβάσει στην επιχειρηματική ελευθερία, γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση, αλλά δυστυχώς όπως σας είπα δεν είναι η βέλτιστη. Τώρα, εάν περιοριστούμε στην μετάδοση για μόνιμη χρήση, δηλαδή έχουμε μια κατάσταση αγοράς και περνάμε βέβαια στο δίκαιο των πωλήσεων. Νομίζω πως ε, βρισκόμαστε στα ανάλογα κεφάλαια της οδηγίας, ε, τα οποία νομίζω μπορούν χωρίς κανένα πρόβλημα να μεταφερθούν και στα του ψηφιακού περιεχομένου και νομίζω πως αυτό ανταποκρίνεται και στην ομοθεσία μεγάλων κρατών μελών όπως της Γαλλίας και της Αγγλίας, κάτι το οποίο δεν νομίζω να είναι καθόλου επίμαχο εδώ πέρα, ότι δηλαδή αυτά ενδείκνυνται να χρησιμοποιηθούν για τον ε, στόχο του ψηφιακού περιεχομένου. Το ίδιο ισχύει βεβαίως ε, και για τα ένομα μέσα νομίζω Βεβαίως ε, δεν ξέρω τι γίνεται με την ε, το δικαίωμα υπαναχώρηση, γιατί και ελαττωματικό να είναι το software, εξακολουθεί, υπάρχει ο πολύ μεγάλος πειρασμός να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί ο καταναλωτής. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην πρόταση της ε, Κομισιόν, βεβαίως αφορά την ρήτρα για περιορισμούς ε, χρήσης ή αντιγραφής γιατί κατά κανόνα εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα που προσανατολίζονται προς τα δικαιώματα του δημιουργού, προς το copyright και πρέπει να μην προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε το copyright από την πίσω πόρτα αν θέλετε, δηλαδή όταν κάποιος αγοράζει έναν υπολογιστή ως καταναλωτής και μετά το χρησιμοποιεί ως επαγγελματίας όπως κάνει ο κάθε φοιτής, να μην ε, έχει προβλήματα με την ομοθεσία του copyright. Επίσης, όσον αφορά το ζήτημα του ε, δικαίου των συμβάσεων, δεν νομίζω πως ε, εφαρμόζεται εδώ πέρα ιδιαίτερα στον τομέα του software. Νομίζω πως η γενική οδηγία ισχύει καλύτερα. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε επί της ουσίας όσον αφορά την εφαρμογή. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Το απλούστερο θα ήταν βεβαίως να γίνει αυτή η παραπομπή στο απτό του πράγματος, να διαγραφεί με αυτή η παραπομπή στο απτό του πράγματος ε, στην οδηγία Βεβαίω ε, πρέπει να είναι σαφές πως αυτό έχει κάποιες συνέπειε. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε ε, έναν κατάλογο εξαιρέσεων γιατί διαφορετικά θα έχει εφαρμογή και σε άλλους ε, Τόμις, ε, όπως ξέρετε, η οδηγία, παραδείγματος χάρη, στα κρυόγραφα κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Επίσης πρέπει να είναι σαφές πως μιλάμε μόνο για την περίπτωση αγοράς, δηλαδή μόνο εκεί πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για εξίσωση με αγαθά στα οποία υπάρχει μια διαρκής χρήση. Μόνο εκεί μπορεί να γίνει παρομοίωση με το software, αν αυτό μεταδίδεται Τώρα το τελευταίο ζήτημα βέβαια ορίζεται θετικά για τον ε, ορισμό κάτι το οποίο βεβαίως μου βάλετε, μου βάλετε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει τολμήσει ένα θετικό ορισμό. Οπότε σημαντικό πρώτα απ' όλα είναι να ξεκαθαρίσουμε πως μιλάμε για ψηφιακά δεδομένα. Επιπλέον να πούμε πως είναι κάτι το μη απτό, κάτι το άειλο, νομίζω αυτό προκύπτει, είναι σαφές. Επιπλέον μιλάμε για ψηφιακά δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται σε αποθηκευτικό μέσο. Διαφορετικά δεν, μπορέσουν, δεν μπορούν καν να αποτελέσουν αντικείμενο κάποιες παροχής εδώ πέρα και η διαφορά ως προς τα αγαθά δεν ε, σχετίζεται με τον τρόπο μεταφοράς. Ανεξαρτήτως δηλαδή του πώς μεταδίδεται αυτό το ψηφιακό δεδομένο. Συνοψίζω. Το δυσκολότερο ερώτημα βεβαίω το οποίο θα πρέπει να κρίνεται είναι το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Θεωρώ πως εξαρτάται πραγματικά από το πως η εμπιστοσύνη έχουμε αν θέλετε στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να το χειριστούν και να το διασφαλίσουν. Τα υπόλοιπα κομμάτια τώρα της οδηγίας, ε, νομίζω πως σύμφωνα και με την εμπειρία των κρατών μελών, μπορούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες να μπορούν να μεταφερθούν και στο ψηφιακό περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed um, ευχαριστώ για τις ξεκάθαρες και ενδιαφέρουσες ιδέες σας δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για να ξεκινήσει τη συζήτηση και για να μας πει αν οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει αντιστοιχούν στο κείμενο αυτό ή αν πρέπει να τις δουλέψουμε περισσότερο. Πριν να δώσω το λόγο στον ε, Ανδρέα Σεβάμπα, Ήθελα και εγώ να καλωσορίσω εδώ για πρώτη φορά τον εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας, την κυρία Κόρτες, που προεδρεύει τη ομάδα Εργασίας για τα Δικαιώματα του Καναλωτή. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας τους επόμενου έξι μήνες και ελπίζουμε να φτάσουμε και συμφωνία με την Προεδρία. Ωραία φιλοδοξία αυτή και επίσης είμαστε πάντοτε ευτυχείς που είναι παρούσα και η Επιτροπή ε, σήμερα εδώ. Ο κύριος Πέτρου θα μιλήσει γι' αυτό αργότερα, αλλά και να καλωσορίσω τον, την, τη νέα διευθύντρια, την κυρία Παρασκευή Μίσου, ε, Μίχου, με συγχωρείτε, ε, που είναι για πρώτη φορά εδώ στην ε, Διευθύντρια της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιτροπής. Ας κάνουμε ένα γύρο συζητήσεων. Λοιπόν, καταρχήν θα πάρει το λόγο ο Ανδρέας Σβάμπ να μας πει τις σκέψεις του για την πρόταση αυτή και τις παρατηρήσεις του για την μελλοντική μας δουλειά, για αυτό το project, καθώς και το πώς προχωρά όσον αφορά τη συγκέντρωση συμβιβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σμιτ Κέσελ και τους και για το ότι μπορέσαμε τόσο πρόθεσμα μέσα στα Χριστούγεννα να συνεννοηθούμε για να σας διαθέσουμε αυτή τη μελέτη και θα ήθελα να σας πω πως έχω πάρα πολύ καλή αίσθηση για την ε, έκθεση αυτή, γιατί νομίζω πως ξεκαθαρίζει πως επί της αρχής το θέμα του ψηφιακού περιεχομένου πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά στα διαφορετικά κεφάλαια της οδηγίας. Την ε, παρουσίαση αυτή την έλαβα εγώ ήδη την Παρασκευή και μπόρεσα να ρίξω μια ματιά και κατέληξα στο συμπέρασμα πως ε, νομίζω πως έχουμε μπροστά μας νέα ζητήματα γιατί συμφωνούμε στο επίπεδο των σκιωδών εισηγητών πως θα θέλουμε να διαγράψουμε τα κεφάλαια 4 και 5 ε, και πρόκειται βεβαίως για τα σημεία εκείνα στα οποία η μελέτη ε, καταλήγει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τη συμπερίληψη, ε, δεν θα αποτελέσουν πλέον αντικείμενο τις οδηγίες μας. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη συγχώνευση των κεφαλαίων 2 και 3 μέσω της ε, συμπερίληψης ε, των κεφαλαίων αυτών. Για να δούμε ποιες ευκαιρίες και κινδύνους αντιμετωπίζουμε. Τώρα, συμφωνώ και πράγματι έχει δίκιο και θέλω να ρωτήσω εδώ πέρα τον κύριο καθηγητή για το εάν συμφωνεί με το ότι οι για το εάν θα πρέπει να αποτελεί χαρακτηρι... Ε, να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα το εάν, ε, για το εάν μπορεί να υπαναχωρήσει κάποιος, το εάν μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον το προϊόν ή την υπηρεσία η οποία του έχει παρισχεθεί και αν αυτό πρέπει να αποτελεί, όπως είπα, τον αποφασιστικό παράγοντα. Θα ήθελα να ακούσω εδώ πέρα την εκτίμηση του κύριου καθηγητή. Αλλά πρέπει να πω πως η Κομισιόν έλεγε μέχρι τώρα πως ε, ε, έχει ζητήσει δύο μελέτες ακριβώς για το ζήτημα της συμπερίληψης του copyright και των δικαιωμάτων του δημιουργού και βεβαίως εάν ε, τα κεφάλαια 4 και 5 δεν θα αποτελέσουν ε, αντικείμενο της έκθεσης, νομίζω πως όλα αυτά μπορούν να λυθούν στο κοινό πλαίσιο αναφοράς. Τώρα βεβαίως αυτό δεν είναι ερώτημα προς τον κύριο καθηγητή, απλά μια παράκληση για περαιτέρω σχόλιο. Βεβαίως επί τη βάση των μελετών, της μελέτης του κυρίου Ροτ έχουμε ήδη ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, αλλά βεβαίως πρέπει να παραδεχτώ πως δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια οριστική κρίση και αξιολόγηση, γιατί εξακολουθώ να ανησυχώ για το εάν και κατά πόσον η επαναχώρηση του καταναλωτή ε, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη από μια τέτοια σύμβαση. Γιατί βεβαίω ο κατασκευαστή αυτού του προϊόντο θέλει να μην συνεχίσει να χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση το προϊόν του. Και αυτό βεβαίω θα μα απασχολήσει εμένα και του χειριστικητέ και αυτή και την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε, σύντομα, κύριε Πρόεδρε, κάποιε γενικέ ε, τοποθετήσει για αυτά τα οποία είπαμε τι τελευταίε εβδομάδε με του χειριστικητέ. Σήμερα είναι η τελευταία δημόσια συνεδρίαση τη Επιτροπή μα πριν από την ψηφοφορία. Γι' αυτό θα ήθελα να φέρω κάποια πραγματάκια τα οποία συζητήσαμε. Συζητήσαμε, δεν αποφασίσαμε. Η κυρία Γκέπχαρτ, βεβαίω η κυρία Τούν δεν είναι εδώ πέρα δυστυχώ σήμερα. Να αναφερθώ λοιπόν σε κάποια από αυτά τα πράγματα. Θεωρώ, αυτή είναι η προσωπική μου εκτύπηση, πως υπάρχει πλειοψηφία για να συγχωνευτούν τα κεφάλαια 2 και 3 στο κεφάλαιο 5 όπου υπάρχει αυτός ο κατάλογος υποχρέωσης πληροφόρησης να δούμε και την σχετική μελέτη των καθηγητών Χάουλ και Ρονχάρτ, οι οποίοι μας είχαν πει πως ε, υπάρχει μια ανάγκη ελάχιστης εναρμόνισης για τις απαιτήσεις υγιεινής ε, και ασφάλειας και νομίζω αυτό θα είναι δυνατόν με τις υποχρεώσεις ε, πληροφόρησης των καταναλωτών. Τώρα, για το άρθρο 12 παράγραφος 4 και το κεφάλαιο 13 θα μπορούν τα κράτη εκείνα τα οποία έχουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας να το διατηρήσουν και στο μέλλον. Επίσης έχουμε βέβαια στο ζήτημα του κεφαλαίου 1 και των υπολείπων των κεφαλαίων 2 και 3 για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στους ορισμούς ιδιαίτερα του email ως ενός διαρκούς ε, μέσου αποθήκευσης. Βεβαίως δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω όλα αυτά εδώ πέρα. Όπως σας είπα, 26 Ιανουαρίου, κύριε Πρόεδρε, έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή και συμφωνούμε με τους ε, σκιώδης Θα το επιβεβαιώσει νομίζω ε, και ο συνάδελφος θα λάβει τώρα το λόγο πως θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα στην ε, ψηφοφορία για να ασχοληθούμε και με τα σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Well, I hope you're right. Uh, ελπίζω να έχετε δίκιο. Συγκητέ, γιατί θα ήταν πολύ καλό να προχωρήσουμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μας ενημερώσατε για το ποια είναι η κατάσταση προόδου. Νομίζω ότι μόνο ο κύριος Ρότσφορ είναι εδώ από τους επίσημους σκιώδεις και θα του δώσω το λόγο και μετά οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση είναι ανοιχτό ο κατάλογος των ομιλητών οπότε πείτε μας αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Εν τω μεταξύ να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόσφορντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο καλύτερες ευχές μου για όλους τους συναδέλφου και συνεργάτες. Ε, θέλω να κάνω, καταρχήν να ευχαριστήσω τον δόκτορα Σμίτ Κέσσελ για την εισηγησή του και θα περιμένουμε να διαβάσουμε και την έκθεσή του. Ωστόσο, να κάνω κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, το ψηφιακό περιεχόμενο είναι ένα μεγάλο τμήμα του μέλλοντος ε, όσον αφορά τις ανταλλαγές και ε, τις καταναλωτικές και άρα τις εσωτερικές αγοράς, γιατί είναι εννοείται ότι η εξαήλωση πολλών στοιχείων και πολλών <laughs> στοιχείων ε, πολλών μάλλον αγαθών είναι στοιχείο αναπόσπαστο της ε, σύγχρονης ζωής και γι' αυτό και πρέπει η οδηγία αυτή που ασχολείται με την κατανάλωση και την κατανάλωση για τα επόμενα 10-20 χρόνια ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να το συμπεριλάβει. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη το ψηφιακό περιεχόμενο. Δεύτερον, το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως και πολλά άλλα στοιχεία κατανάλωσης, θα γίνουν ε, όλο ένα και περισσότερο αντικείμενο εξ αγορών. Το ψηφιακό περιεχόμενο συχνά το αγοράζουμε εξ Όλα τα αγοράζουμε όλο ένα και περισσότερο εξ και το ανέφερε αυτό και ο Δόκτωρ Σμιτ και είναι σαφές και η ομάδα μου θεωρεί πως η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή κυρίως είναι χρήσιμη εφόσον ασχολείται με την ανάπτυξη των εξαποστάσεων αγορών. Έπειτα, το δικαίωμα αυτό εκμετάλλευση είναι το βασικό, το δικαίωμα επαναχώρηση είναι το βασικό πυλώνα ε, για τι αγορές εξαποστάσεως. Το θέμα λοιπόν το πιο σημαντικό που πρέπει να ρυθμιστεί είναι πώς θα καταστεί συμβατή η συναλλαγή για το ψηφιακό περιεχόμενο με το δικαίωμα επαναχώρηση. Αν δεν βρούμε λύση για αυτό το πρόβλημα θα είναι δραματική κατάσταση, γιατί αυτό θα αφισβητήσει το ίδιο το κέντρο βάρους της οδηγίας που εφόσον αφορά τις εξαποστάσεις αγορά, αγορές είναι το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Μιλήσατε για τα παιδιά σας, μπορούμε να μιλήσουμε όλοι για τα παιδιά μας. Όλοι γνωρίζουμε πόσο εύκολο είναι να αγοράσεις και να ε, παραγγείλεις διάφορα ε, προϊόντα ψηφιακού χαρακτήρα και γι' αυτό και πρέπει αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Έπειτα, θα πρέπει και να θέσουμε τι επιχειρήσει ενώπιον των ευθυνών του ω προ αυτό. Δηλαδή, επιχειρήσει που πουλούν ψηφιακό περιεχόμενο. Θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και αυτές, να δουν πώς δηλαδή θα κατασκευάσουν το προϊόν τους. Γιατί πρόκειται για προϊόν το οποίο είναι άειλο αλλά είναι προϊόν. Πώς λοιπόν θα το κατασκευάσουν έτσι ώστε να είναι συμβατό με το δικαίωμα επαναχώρησης. Πώς δηλαδή θα καταφέρουμε τα προϊόντα αυτά ακόμα και αν τα ανοίξει κανείς, ακόμα και αν ε, μπορούν να, μπορεί κανείς να τα αντιγράψει, ε, να είναι προστατευμένα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα της επαναχώρησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Από ό,τι κατάλαβα αυτό σκέφτεστε κι εσείς και συμφωνώ απόλυτα. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε κάποιες παρατηρήσεις γιατί ο εισηγητής ε, στα όσα είπε κάπως διέβαινε τη συζήτηση για να μας εξηγήσει την κατάσταση προόδου του θέματος. Συμφωνώ με τα όσα είπε, είναι πολύ σημαντική δουλειά. Ο κύριος Σβάμπ κινητοποιεί ολόκληρη την ομάδα του, το επιτελείο του, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτές τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Πολλά πράγματα, όπως είπατε, Πρόεδρε, βέβαια πρέπει ακόμα να τα εξετάσουμε. Δεν θέλω να επανέλθω. Είμαστε υπέρ της συγχώνευσης των κεφαλαίων 2 και 3. Ε, να θυμίσω απλά ότι, και είναι ένα σημαντικό θέμα για την ομάδα μας, ότι έχουμε μια πολύ ρεαλιστική άποψη όσον αφορά αυτή την οδηγία και ένα συστημικό ζήτημα είναι ότι όσο το σκέφτομαι, τόσο λιγότερο πιστεύω πω η οδηγία αυτή θα λύσει όλα τα προβλήματα του καταναλωτή για τα επόμενα 20 χρόνια. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο ρεαλιστικοί, να επιστιάσουμε την προσοχή στα πιο σημαντικά ζητήματα και εδώ στη συγχώνευση του 2 και του 3 να πούμε ότι για τις εξαποστάσεις αγορά, αγορές ή εκτός ε, ε, χώρου πωλήσεων αγορές. Αυτό, αυτό είναι το θέμα το πιο σημαντικό, αυτό πρέπει να λύσουμε. δεν πρόκειται για συμβασμό με το Συμβούλιο ή ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε το Συμβούλιο. Όχι, είναι η δική μα άποψη αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε συμβαστικέ λύσει για τα κεφάλαια 4 και 5. Μπορούμε κάλλιστα να περιοριστούμε σε μια οδηγία που θα εστιάζει την προστοχή στα κεφάλαια 1, 2, 3 και να θέσουμε λίγο στην άκρη τα 4 και 5 και οι επόμενε οδηγίε που θα ρυθμίζουν αυτά τα θέματα να είναι εφαρμοστές. Φυσικά να πω και δύο λόγια γιατί ο Ανδρέας αναφέρθηκε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή που πλησιάζει σε δύο, δυόμιση εβδομάδες νομίζω εδώ θέλω να πω και ίσω είναι κάπω προσωπική άποψή μου, αλλά η Ευρώπη σήμερα δεν πάει καλά. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και στους πολίτες της είναι δύσκολε. και γι' αυτό και πρέπει να το πούμε και εδώ, όσο γίνεται περισσότερο στην Επιτροπή μας, να φτάσουμε σε μια συνενετική, ένα συνενετικό κείμενο για αυτά τα θέματα του καταναλωτή. Καλύτερα λιγότερα πράγματα, αλλά να συμφωνούμε όλοι, ε, μπορεί να μην τροφοδοτήσουμε δηλαδή μια συζήτηση τεταμένη. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη ε, για ένα θέμα τόσο σημαντικό η κατανάλωση, που όπως γνωρίζετε είναι ένας ε, βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε την ανάπτυξη, ο καταναλωτής είναι ανήσυχος, ο Ευρωπαίος καταναλωτής ανησυχεί όσον αφορά την οικονομική κρίση και τα προγράμματα ανάκαμψης στις διάφορες χώρες. Πρέπει να βρούμε δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο να τον καθησυχάζει και όχι να τον ε, ε, από προσανατολίζει να, τον, να δημιουργεί περισσότερη αστάθεια. Αυτά, Πρόεδρε, ήθελα να κάνω αυτά τα σχόλια και πάλι να σας ευχαριστήσω για αυτή τη ε, δουλειά του κυρίου Σμιτ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Ροσφόρ για την ε, συμβολή σας στη συζήτηση και την όλη ανάλυση του θέματος αυτού. Δεν ε, έχω στον κατάλογο μιλητών κάποιον άλλο ε, συνάδελφο μέχρι στιγμής. Θα παρακαλέσω λοιπόν πρώτα απ' όλα την Επιτροπή να ακούσουμε κάποια σχόλια σε σχέση με όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα και στη συνέχεια την εκπρόσωπο του Συμβουλίου εφόσον το επιθυμεί. Κύριε Πέτρη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να ε, πω και εγώ κάποια πράγματα σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση και βέβαια συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο και το ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο παρουσίασε σήμερα ο καθηγητής Σμιτ Κέσελ. Λοιπόν, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία περί δικαιωμάτων των καταναλωτών πράγματι κάλυπτε τις ψηφιακές υπηρεσίες ε, και στο ψηφιακό περιεχόμενο σε, ως ένα βαθμό θα έλεγα ε, συμβάσεις ε, εξ αποστάσεως ή εκτός χώρων πωλήσεως. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά τους κανόνες για αθέμητους όρους αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τις συμβάσεις αγοραπολισίας εκτός εγκαταστάσεων πώλησης κτλ. Είναι ενδιαφέρουσε οι σκέψει του συντάκτου ενημερωτικού εγγράφου, ο οποίο ε, επισημαίνει κάποιε σημαντικέ πτυχέ. Είναι σαφέ ότι ο καταναλωτής πρέπει να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο προτού το μεταφορτώσει, προτού το κατεβάσει, επί παραδείγματα. Και αυτό προβλέπει και η πρόταση άλλωστε. Πιο δύσκολο βέβαια είναι το ζήτημα της παναχώρησης. Αν θα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα ο καταναλωτής σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο. Εδώ η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εξή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ε, του καταναλωτή εκπνέει, πάβει να ισχύει από τη στιγμή που ξεκινήσει τη διαδικασία μεταφόρτωσης. Έχει δηλαδή ο καταναλωτής δικαίωμα υπαναχώρησης αφού συνάψει τη σύμβαση, αν αυτό γίνει επιγραμμικά, online, πριν όμως ξεκινήσει τη μεταφόρτωση. Η διάκριση αυτή παραμένει στο κείμενο. στο κείμενο για το οποίο υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη γενική προσέγγιση. Και υπάρχει και ειδική παρέκκληση σε ό,τι αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο που αρχίζει να ισχύει άμα την ανάρξη της ε, μεταφόρτωσης. Αυτό είναι μια βελτίωση στο κείμενο της Κομισιόν και θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, εάν μιλάμε για μια κατάσταση όπου αποτέλεσμα της σύμβασης, της οδηγίας, συγγνώμη, για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι να επικεντρωθεί σε αυτό που προτείνει το Κοινοβούλιο, δηλαδή στις εξαποστάσεως ή εκτός χώρων πολίσεως συμβάσεις, τότε το κείμενο ως έχει, κατά την άποψή μας, νομίζουμε ότι προστατεύει, εξασφαλίζει επαρκή προστασία για τον καταναλωτή και αντιμετωπίσει και τα ζητήματα του ψηφιακού περιεχομένου με επαρκή τρόπο. Ποιο είναι όμως το επίμαχο ζήτημα που έχει τεθεί και αλλού. Είναι το θέμα της συμμόρφωσης των αγαθών αυτών ε, με τις συμβάσεις. Κεφάλαιο 4 δηλαδή. Και αν υπάρχουν ένδικα μέσα σε περίπτωση που δεν είναι ε, επαρκές ή είναι λεπτοματικό το περιεχόμενο. Κατά την άποψή μας είναι ιδιαίτερα ε, πολύπλοκο το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι και το ενημερωτικό έγγραφο το επιβεβαιώνει αυτό. Ιδίω λόγω του ε, ότι είναι δύσκολο να οριστεί το ψηφιακό περιεχόμενο αλλά ε, και η εφαρμογή των ένδικων μέσων. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει περαιτέρω το όλο ζήτημα και ανέθεσε ε, δύο εκθέσεις να γίνουν. Η μία θα αφορά τα οικονομικά ζητήματα και το κατά πόσον υπάρχει ζημία για τον καταναλωτή. Χρειάζεται να ρυθμιστεί δηλαδή το θέμα αυτό. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη. Και η δεύτερη είναι το να δούμε τα νομικά ε, στοιχεία. Να δούμε την ομολογία, την ομοθεσία των κρατών μελών, για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο το ψηφιακό περιεχόμενο. Εδώ βλέπουμε ε, τα αποτελέσματα, μάλλον περιμένουμε τα αποτελέσματα εντός του έτους και μάλλον θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα τον Ιούνιο. Οπότε ελπίζουμε τότε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης και τις ανάγκες να αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό περιεχόμενο πιο διεξοδικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας ε, για τους καταναλωτές. Κάτι που ανέφερε και ο κύριος Φάπ τώρα. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε και για το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο τα σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο. Ε, νομίζω ότι είναι καλό θα δούμε και ποια θα είναι εκβάση των συζητήσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και αν αυτό θα οδηγήσει σε μια οδηγία η οποία θα εστιάζει στις εξαποστάσεως ε, συμβάσεις ή εκτός ε, πρατηρίων, εκτός καταστημάτων ε, συμβάσεις off-premises στα αγγλικά. Και ίσως καλό θα ήταν να δούμε και πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα πορίσματα των μελετών που έχουμε αναθέσει στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι ο εισηγητής, ο κύριος Σβάπ, φαίνεται να είναι ευνοϊκά διακείμενος σε ό,τι αφορά την πορεία, την κατεύθυνση των εργασιών στο Συμβούλιο και από ό,τι φαίνεται συμμερίζεται την ε, άποψη αυτή και ο κύριος Ροσφόρ. Και βέβαια και εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε θετικά, ατενίζουμε θετικά και το, μέλος, το μέλλον συγγνώμη, των διαπραγματεύσεων σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την αρχή σας αυτή απάντηση. Φαντάζομαι ότι είναι προφανές ότι πολλά είναι τα στήματα που χρήζουν εξέτασης. για το κοινό πλαίσιο δεν έχουμε νομίζω συμφωνήσει. Ακόμη πόρο απέχουμε, θα το δούμε και αργότερα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αφήσουμε να περιμένουν τόσο καιρό οι καταναλωτές, βέβαια θα το δούμε. Κυρία Κέτες από τη Συμβουλή θα ήθελε ίσως πρώτα απ' όλα να μας συστηθεί και μετά να μας πει και κάποια πράγματα για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στο Συμβούλιο. Ε, κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος της Προεδρίας της Ουγγρικής σας καλωσορίζω σε αυτή την συνεδρίαση. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι υποδομητική η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η μέχρι στιγμή πείρα δείχνει πως δεν θα έχουμε προβλήματα. Πάντα συνεργαζόμασταν με ευκολία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα όσον αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, το Συμβούλιο έχει μια πρώτη θέση η οποία ευθύθηκε στην Κορεπέρ αλλά χρειάζεται ακόμα γύρω στις 15 μέρες θα έλεγα για να οριστικοποιηθεί αυτή η θέση και να υιοθετηθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου του Συμβουλίου των Υπουργών. Αυτό θα γίνει σύντομα. Και η Ουγγρική Προεδρία βέβαια θέλει να σημειώσει όσο δυνατόν περισσότερη πρόοδο με τις διαπραγματεύσεις και θα θέλαμε να συνεργαστούμε στενά και με, το Κομισιόν, με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα τις διατάξεις για το ψηφιακό περιεχόμενο, καλωσορίζουμε την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις ε, των ειδικών και των βουλευτών. Σύμφωνα δε με την ε, προκαταρκτική θέση του Συμβουλίου δεν εμπίπτει σε αυτούς τους κανόνες το ψηφιακό περιεχόμενο γιατί δεν είναι ούτε αγαθά ούτε υπηρεσίε, Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε αργότερα στο Συμβούλιο. Οπότε πρέπει να επαναλάβω εδώ πέρα πώς βασιζόμαστε στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί σας και θα θέλαμε να συνεχίσουμε βεβαίω την καλή δουλειά που έχουμε ξεκινήσει επί Βελγικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και αναμένουμε και εμείς να σας δεχτούμε ξανά στην Επιτροπή μας και να σημειώσουμε πρόοδο. Να ευχαριστήσω βεβαίως και τη Βελγική Προεδρία για τις προσπάθειές της σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούσαμε Συμβούλιο και Κομισιόν. Θα έδινα τον λόγο στον Άντριου Σβάμπ. Απλά δεν ξέρω αν και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Σμιτ Κέσελ θέλει να επανέλθει, να απαντήσει στα σχόλια τα οποία ακούστηκαν. Δύο λόγια, ναι βεβαίως. Υπάρχουν, όσον αφορά το δικαίωμα επαναχώρησης, κάποιες, κάποιες, ενδιάμεσες, κάποιες ενδιάμεσες οδοί, τις οποίες μπορούμε να δούμε, που σημαίνουν πως ε, δεν θα αποκλείεται το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά θα προσπαθήσουμε ε, να το αντισταθμίσουμε μέσω κάποιου είδου αντικατάστασης ή αποζημίωσης. Και φαινώς αυτό είναι δυνατόν και είναι και η ισχύουσα γερμανική λύση. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια μέση οδό εκεί πέρα, δηλαδή να εξαρτάται από κάποιες επιπλέον πληροφορίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί εκ των προτέρων και στην περίπτωση που δεν είχαν παρασκευθεί αυτές οι πληροφορίες. Δεν υπάρχει πλέον απέτηση σε τέτοιο δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν δεν είχε γίνει αυτό λοιπόν, ε, χάνονται. Αυτή είναι η γερμανική συζήτηση θα έλεγα, η οποία έχει δείξει πως πάντα είναι καλύτερο τέτοια ζητήματα να ρυθμιστούν στην ε, πλευρά των ε, ένομων συνεπειών παρά από την πλευρά των προϋποθέσεων της ε, σύμβασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ βεβαίω και για το φάκελο τον οποίο προετοιμάσατε. Λυπούμε που δεν μπορέσαμε να δώσουμε αντίγραφα σε όλου. Νομίζω πω θα είναι διαθέσιμα όλα αυτά την Τετάρτη και θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πριν καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση. Νομίζω πως ε, είχατε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ακόμα και αν δεν ενσωματωθούν σε αυτό το πρώτο πακέτο. Ε, κάτι το οποίο βεβαίω θα ξαναδεί, φαντάζομαι, ο εισηγητής Άντριου Σφαμπ θα ήθελε να συνοψίσει για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ή τίποτα άλλο που θα ήθελε να πει στην Επιτροπή μας. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε έχει πάει πέντε παρά με Λοιπόν, βλέπετε τα θέματα τα οποία έθεσε ο κύριος καθηγητής, τα οποία θα πρέπει να δούμε. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ροσφόρ, πως ειδικά για τους νέους καταναλωτές είναι ένα σημαντικό σημάδι αυτό για το ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε κάτι μόνο εάν μπορούμε να το κάνουμε σε μια στέρεη, στιβαρή νομική βάση. Αλλά κύριε Πρόεδρε, σας διαβεβαιώνω πως... Ε, και αυτό και τα άλλα ζητήματα θα τα δούμε με την απαιτούμενη πρόσοχη και στις 26 Ιανουαρίου θα έχουμε να προτείνουμε μια κατάλληλη συμβαστική λύση. Τίποτα άλλο δεν έχουμε πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Right. Well, thank, I'd like to thank everybody very much. Just... Να σας ευχαριστήσω όλους. Να επιβεβαιώσω ότι θα ψηφίσουμε στις 26 Ιανουαρίου στις 3 ε, για, αυτό το, για αυτή την πρόταση και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει πολλή δουλειά με τον εισηγητή και τους σκιώδης πριν από εκείνη την ημερομηνία. Πριν να κλείσουμε θέλω να, να γνωρίσω τον να ευχαριστήσω τον Άντριου Στέγγινς που είναι τελευταία φορά εδώ. Έχει αλλάξει επιτροπή. Επιτροπή ασφάλειας και άμυνας. Εκεί θα πάει τώρα ε, λόγω εξέλιξης της διαδρομής. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του στην Επιτροπή μας και ιδιαίτερα διότι φρόντισε για το θέμα των, δικαιωμάτων του καταναλωτή και να καλωσερίσω και τον νέο υπάλληλο που θα αναλάβει τη θέση του. Λοιπόν, είναι λίγο πριν τις 4, σύντομο διάλειμμα για όσους δεν θέλουν να μείνουν για την ψηφοφορία στις 4, αλλά και για να μπορέσουν οι πολιτικές ε, ομάδες να καλέσουν ε, τους συναδέλφους. Θα αρχίσουμε λοιπόν στις 4 ακριβώς. Uh, so, ladies Συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Τη συνεδρίασή μας αυτή, την πρώτη για το 2011. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να θέσω σε ψηφοφορία την ε, τελική θέση, τη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση που επιβεβαιώνει και την έκβαση των διαπραγματεύσεων των οποίων ηγήθηκε η συγκήτριά μας ε, Κάθριν Στάιλερ με τη Βελγική Προεδρία. Το πλήρες κείμενο της πρότασης έχει διανεμηθεί, το έχουν μελετήσει οι σκιώδεις εισηγητές. Ήταν πολύ αποτελεσματικές οι διαπραγματεύσεις τον οποίο προείδευσα και μετά από υπόδειξη των σχεδόν έγραψα επιστολή στον κύριο Φαν Κουίκεμπορν, το Βέλγο Υπουργό που τον γνωρίζετε φαντάζομαι και τον ευχαρίστησα για την ε, συνεργασία του. Ζήτησα επίσης να μας δώσει η Προεδρία μια σαφή εξήγηση για το γεγονός ότι αρκετά αργά πρόσθεσα μια εντελώ καινούργια παράγραφο. Δέχθηκαν βέβαια οι συγγητές να συμπεριληφθεί η παράγραφος αυτή. Προς ενημέρωσή σας να σας πω απλά ότι στη συμφωνία οι 60 από 83 τροπολογίες που είχαμε εγκρίνει στη συνεδρίασή μας στις 22 του έγιναν δεκτές. Βλέπετε λοιπόν πόσο καλά τα πήγε η διαπραγματευτική μας ομάδα υπό την κυρία Στάιλερ. Θέλω πρώτα να παρακαλέσω τους κοιότητες συζητητές αν θέλουν να πούν κάτι. Όχι. Α, η κυρία, η Ρούλη. Η κυρία Ρούλη θέλει να πει κάτι. Και αντιπρόεδρος μας. herr liebe kolleginnen und kollegen meine damen und herren! Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πράγματι, οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι, stakeholders όπως ε, τους λέμε, μας έδωσαν αρκετές πληροφορίες. Κάποιες φορές ε, με κάποια καθυστέρηση βέβαια, αλλά μεταξύ της εισηγήτριας ε, σκιωδών εισηγητών και με τη συνεργασία και των ε, υπόλοιπων θεσμικών οργάνων νομίζω ότι καταφέραμε να φτάσουμε στην ε, συμβιβαστική αυτή πρόταση. Φυσικά ο συμβιβασμός δεν είναι κάτι που αφήνει τους πάντες ικανοποιημένους, άρα ούτε και εμένα, αλλά έχουμε αυτό το συμβιβασμό και νομίζω ότι το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη λεγόμενη διαδικασία της Επιτροπής όπως την ε, αποκαλούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να δουλέψει και εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω το συντομότερο δυνατό, θα πρέπει να συνεργαστεί με την εισηγήτρια, με τους σκιώδεις εισηγητές, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία λύση σε σχέση με τα αναπάντητα μέχρι στιγμής ε, ερωτήματα. Και νομίζω ότι θα γίνει αυτό, ελπίζω τουλάχιστον να γίνει αυτό και με αυτές τις παρατηρήσεις προτείνω και εγώ τώρα να περάσουμε σε ψηφοφορία. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρούλε. Θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την επιστολή την οποία στείλατε στη Βελγική Προεδρία. Πιστεύω ότι διαφορετικά η τροπολογία που κατέθεσα δεν θα είχε γίνει δεκτή. Χάρη στην επιστολή που στείλατε κύριε Πρόεδρε μπορούμε ως πολιτική ομάδα να δεχθούμε το συμβεβαστικό κείμενο. Συμφωνώ και με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Μάγερ, ότι τώρα πρέπει να δούμε πώς θα μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο ο κανονισμός αυτός. Και όπως συχνά συμβαίνει με τους συμβιβασμούς, ε, υπάρχουν κάποια στήματα που έχουν μείνει αδιευκρίνιστα. Επευθύνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ώστε να έχουμε μια μελλοντική συνεργασία που θα δώσει ένα πολύ ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα. Κάτι σας είπα και για τον Βέλγο Υπουδρό και σας είπα ότι ζήτησα να υπάρξει μια διευκρίνηση στη συζήτηση ε, που θα έχουμε στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Οπότε και τότε και εσείς κυρία Ρούλε μπορείτε να λάβετε το λόγο και να πείτε αυτά που θέλετε. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κανόνες εφαρμογής και τη διαδικασία εφαρμογής φαντάζομαι ότι θα σημειώνουν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν αυτά που είπατε. Βλέπω ότι υπάρχουν και νεύουν μάλιστα. Και αν θέλει και Επιτροπή το λόγο σίγουρα θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Δεν ήθελα να έχουμε μια γενική συζήτηση, αλλά και η αντιπρόεδρος μας, κυρία Βερνιό, θέλει κάτι να πει. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να πω απλά ότι η κυρία Στάιλερ, η Κατρίν ε, δεν είναι εδώ. Μου ζήτησε να μιλήσω αντί αυτής. Δυστυχώς δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν δύο προλαλήσαντες, αλλά και η Κάθριν το ίδιο ακριβώς μήνυμα ε, ήθελε να διαβιβάσει εδώ. Πάντα υπάρχουν ε, στους συμβιβασμούς κάποια σημεία που μας αφήνουν ανικανόπιτους, αλλά νομίζω ότι όλοι μαζί ε, τα καταφέραν πολύ καλά και η Κάθριν Διεμού ήθελε να σας ευχαριστήσει όλες και όλους για την πολύ επικοδομητική αυτή συνεργασία, ιδίως για αυτόν τον δύσκολο, τον δύσκολο συμβιβασμό που πετύχαμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι εκπροσωπούσε την κυρία αλλά θα σου είχα δώσει αμέσω το λόγο. Η Επιτροπή θέλει να σχολιάσει συντόμω Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και την κυρία Στάιλερ και τους κοιόδης εισηγητές για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο επιτελέσατε στην συνεδρία του τριμερούς διαλόγου. μιση ώρες διήρκεσε αυτή η συνάντηση και νομίζω ότι χάρη σε αυτήν τη συνάντηση επιτύχαμε το συμβιβασμό. Και εμεί το ίδιο θεωρούμε. Ο συμβιβασμό είναι συμβιβασμό. Άρα δεν είναι πλήρω ε, ικανοποιητικό ε, για κανέναν, αλλά είναι σημαντικό παρόλα αυτά ο συμβιβασμό που πετύχατε με το Συμβούλιο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια πάντοτε είναι πρόθυμη να συνεργάζεται με τους ηγητές, με τους σκιώδες ηγητές, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό βέβαια και φυσικά και είμαστε πρόθυμοι να επιταχύνουμε τις εργασίες ό,τι αφορά τις κατεξοδότηση πράξη. Δεν ξέρω ακριβώς ε, πού αναφέρονταν οι σκιώδες ηγητές. Ε, βέβαια, ήδη έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες με τους stakeholders που είπατε και εσείς, με τους ενδιαφερομένους ε, φορείς και φαντάζομαι ότι θα επιταχυνθεί και η όλη διαδικασία με την κατεξιοδότηση ε, πράξη, αλλά νομίζω ότι ε, αυτό ε, που προβλέπουν και οι κανονισμοί θα είναι λίγο πολύ το διάστημα των δύο ετών. Δεν νομίζω νωρίτερα από δύο χρόνια δηλαδή. Να έχουμε κάποια εξέλιξη. Φυσικά θα συνεργαστούμε με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο και θα διατηρήσουμε τις επαφές που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Um, επειδή παρίσταται και η Βελική Προεδρία, θα διαβιβάσω και σε αυτούς τις ευχαριστίες. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε μετά την ψηφοφορία. Να στείλουμε μία επιστολή στην Κομισιόν με κάποια ζητήματα και να σας παρακαλέσουμε να μας ε, διαβιβάσετε ένα non-paper, μια μικρή έκθεση για το πώς ε, βαίνει η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα ήθελα να θέσω σε ψηφοφορία, ε, με μία ενιαία ψηφοφορία το πακέτο αυτό. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά υπάρχουν. Εγκρίνεται ομόφωνα. Έχουμε και τους αριθμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια θα συγχαρούμε την κυρία Στάιλερ που λόγω των χιονοπτώσεων έμεινε στη Σκοτία δυστυχώς. Κόλλησε εκεί, δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και η συζήτηση νομίζω έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα ή την Τρίτη. Α, Δευτέρα, Δευτέρα 5 και 4 το απόγευμα στην επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούρτου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία, έκθεση της κυρίας ε, Μακλάρκιν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χαρά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια να κάνει μια εισαγωγή πριν την ψηφοφορία και από ό,τι είδα ε, το ΕΛΚΑ θέλει να προτείνει κάποιες καθυστερημένες προφορικές τροπολογίες. Δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε. Καλό θα ήταν να μας το πείτε, αν δέχεστε πάντως αυτές τις προφορικές τροπολογίες. Και για ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για την βοήθειά τους και την συνεργασία τους, ιδιαίτερα δεδομένου του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που είχαμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω πως η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς μπορεί να συμβάλλει σημαντικά μέσω αυτής της γνωμοδότησης για την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος να αναγνωρίζουμε ότι οι ανισότητες στην υγεία βασικά οφείλονται στις, ε, σε κοινωνικο-οικονομικούς ε, λόγους, αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τη ε, πτυχία που ισχύουν στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να χαίρει ο τομέα αυτό τη ίδια ε, ελευθερία κυκλοφορία, κυκλοφορία, αλλά λόγω τη ιδιαιτερότητα τη δουλειά αυτή θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλε δικλείδε ασφαλή, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ε, εργασία κατάλληλων ατόμων στον τομέα. Και γι' αυτό και είναι και η Κομισιόν εδώ για να ασχοληθεί με το θέμα των επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα του ελέγχου των επαγγελματικών προσόντων. Όσον αφορά τις προφορικές τροπολογίες που πρότεινε το ΕΛΚ, τις έχω δει και τις εγκρίνω. Ευχαριστώ. Thank you very much else? Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο να σχολιάσει πριν ψηφίσουμε. Ωραία. Να ελέγξω. Α, κυρία Βερνιό. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΜΑ που αρμονικά συνεργάστηκε μαζί μας για ένα θέμα τόσο ευρύ και περίπλοκο αλλά πιστεύω πως θα μπορέσουμε να δώσουμε μια γνωμοδότηση αρκετά εναρμονισμένη και ισορροπημένη για την Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος και θέλω να πω ότι οι τροπολογίες του ΕΛΚ δεδομένου ιδιαίτερα στις 44 είχαμε ε, αρχικά σκεφτεί να καταψηφίσουμε για μια συγκεκριμένη λέξη που είχε δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όμως εφόσον η τροπολογία αυτή έχει διορθωθεί, θα υπερψηφίσουμε τις 44. Ευχαριστώ. κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ε, ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους και σε εσά Πρόεδρε και να πω σύντομα ότι εκτιμάμε στο ΕΛΚ την θέση της ε, εισηγήτριας και την ευχαριστούμε για το πνεύμα συνεργασίας που έδειξε, δέχτηκε τις τελικές μας τροπολογίες μέσα στη μέση των γιορτών, ε, επεξηγώνται αυτές και στον κατάλογο ψηφοφορίας και για να σας πω ότι αυτή η γνωμοδότηση ε, θα συμβάλλει πάλι σοβαρά ώστε σε μια εποχή κρίσης να περιοριστούν οι ανισότητες στην υγεία στο πλαίσιο της πολιτικής υγείας του κάθε ε, κράτους μέλους. Σας ευχαριστώ. Right. Άλλος και όδης. Uh, Όχι. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να ελέγξουμε αν όλοι έχετε τις κάρτες σας. Ε, να κάνουμε το συνηθισμένο έλεγχο, γιατί έχουμε αρκετές ψηφοφορίες. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε. Ας ψηφίσουμε πρώτα ε, τα μέλη του ΕΛΚ. Uh, we have 11 for the EPP. Should be 13, so you're 200 at the moment. The vote is closed for the EPP. Τέλος της ψηφοφορίας. We'll record you separately then. Uh, S&D. Οι σοσιαλιστές να ψηφίσουν τώρα. S&D, the vote is open. Η κυρία Βερνιά έχει ξεχάσει την κάρτα της, οπότε θα την, μετράμε χωριστά. Πέντε μόνο. Έξι, οπτά. I'll count you manually Εντάξει, σας θα σας μετράω χωριστά και νομίζω όλους τους υπόλοιπους σας βλέπω. Εντάξει, έχουμε τέσσερις φιλελεύθερους, τρεις ECR ε, και δύο πράσινους. Και έχουμε τον Τένις από την ΚΟΥΕ, την κυρία Στάσερ. Ωραία, ξεκινάμε. Ψηφίζουμε λοιπόν καταρχήν τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σχεδόν ομόφωνα. Οπότε προχωράμε στην τροπολογία 4 για την παράγραφο 1α νέο από τον κύριο Ζουβά υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 Μακλάρκιν υπέρ κατά εγκρίνεται. We then move to compromise amendment 2. Those in favor. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και προχωρώμε στην τροπολογία 6 της κυρίας Μπάστος. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Βερνιό, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Παρβανόβα. Υπέρ εδώ α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψηφίζουμε λοιπόν για τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. And Mrs. Vanier is poor. Uh, the vote is closed. Uh, so it was four... Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κυρία Σάλντε Μόζε, τροπολογία 8. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 8. Σολτεμόζε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 κατά. Περνάμε στην τροπολογία 11. Βερνιό. Υπέρ. Ας ψηφίσουμε. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 3, συμβαστική 3, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 18, την κυρία Σαλντεμόζ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, Μακλάρκιν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Μακλάρκιν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Βερνιό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Εδώ νομίζω πως έχουμε μια προφορική τροπολογία για την 22. Η κυρία Μπάστος θα μας τη διαβάσει για τα πρακτικά. Μπορείτε να μας τη διαβάσετε παρακαλώ. Αντικαθιστά την... Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τροπολογία αφορά τη διαγραφή των λέξεων and remuneration. Actually on the voting list, I think. Μάλιστα. Λοιπόν, τροπολογία του κύριου Ζουβέν, λοιπόν, με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24, Βερνιό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. In favor. The So that's uh, Defeated. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 17 κατά. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 Μακλάρκιν. Επόμενη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 Γκρέχ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Γκρέχ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 30. The vote is Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 20 κατά 1 υπέρ. 10 υπέρ, συγγνώμη. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και περνάμε έτσι στην τροπολογία 35 της κυρίας Μακλάρκιν για την παράγραφο 5α. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Παρβανόβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Ζουβά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Βερνιό. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 37 της κυρίας Βερνιό. Εγκρίνεται. 16 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Παράγραφος 6. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 42 Παραβανόβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 43, προφορική τροπολογία. Είναι η ίδια όπως αυτή που έχουμε στον κατάλογο ψηφοφορίας. Είναι η ίδια, μάλιστα. Είναι στον κατάλογο ψηφοφορίας λοιπόν και ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία 43. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 44 της κυρίας Μπάστος. Και εδώ είναι ο κατάλογο ψηφοφορίας, οπότε ας ψηφίσουμε 44 όπως έχει διδοποποιηθεί, υπέρ, κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται, μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Γιατί 44. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21, 21 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 45. Μπάστος. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 45. Vote 22. Εγκρίνεται με 22 ψήφου υπέρ. Συμβιβαστική 7 τώρα, στην παράγραφο 7 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επομένως, περνάμε στην τροπολογία 49, τροπολογία Ρούλε. Ψήφι υπέρ. Μάλλον, ας α, ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι, συγγνώμη. Θα πάω, Γιατί να πάμε στην 51, εγώ νομίζω στη 49 πρέπει να πάμε. 49 λοιπόν. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 ψήφι υπέρ, 20 κατά. Τροπολογία 46, Μέλτσερ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 46. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται με την ίδια αντιστοιχεία ψήφων, 10 υπέρ, 20 κατά. Τροπολογία 51, Μακκλάρκιν υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 52 μπάστος, ψήφι υπέρ, κατά. Ας το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 52 μπάστος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται η τροπολογία 52, 22 προς 8. Τροπολογία 53 μπάστος, ψήφι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 Βερνιό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 Μπάστος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 56 Μπάστος υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Εδώ ολοκληρώνουμε την ψηφοφορία επί των τροπολογιών και ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 28 ψήφι υπέρ, 2 κατά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και συγχαρητήρια κυρία Μακλάρκιν. Και είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσετε η Επιτροπή Περιβάλλοντος να λάβει υπόψη τις ε, πολύ σημαντικές και πρακτικές υποδείξεις της Επιτροπής μας. Και τώρα Περνάμε στην γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ενέργειας για την έκθεση πρωτοβουλίας με θέμα τη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ε, είναι ο κύριος Κρόιτσμαν, εισηγητής, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω βέβαια να ευχαριστήσω και τους ε, εισηγητές από τις ε, λοιπές πολιτικές ομάδες Προσπάθησα να εστιάσω σε πτυχές που δεν κάλυπτε η έκθεση ΛΑΝ και βέβαια υπήρξε μια σειρά τροπολογιών που πήγαν πιο πέρα από αυτό το πεδίο. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες για τις οποίες δεν έχω καμία αντίρρηση και γενικώ προσπάθησα να προτείνω συμβαστικές τροπολογίες ε, Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που αφορούν ε, κάποια σχέδια πολύ σημαντικά όπως τον Γαλιλαίο για παράδειγμα με δισεκατομμύρια ε, για ποσά εκεί κάπου ε, είμαι λίγο πιο προσεκτικό στην τοποθέτησή μου αλλά γενικώ σας ευχαριστήσω όλους όσοι έχουν συνεργαστεί και να μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε λοιπόν απευθεία στην ψηφοφορία και ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 1, στην παράγραφο 1. Ψήφι υπέρ. Υπάρχουν ψήφι κατά. Ε, άρα συντριπτική είναι αυτή που ψήφουν υπέρ, η πλειοψηφία λοιπόν. Τροπολογία 2 από κάποιους συναδέλφους, ε, ψήφι υπέρ, κατά Αποχές υπάρχουν. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Όλο το κείμενο εκτός από τις λέξεις «anotomatic». Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, ψήφι περ. Κατά. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, δηλαδή τις δύο λέξεις που προανέφερα, ενατομάτικ. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 20 ψήφοι κατά και 10 υπέρ. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 4, που επίσης χωρίζεται σε τμήματα, όπως βλέπετε και στην, στο χαρτί που έχετε μπροστά σας. Δεν θα σας αναγνώσω τα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 2α, τροπολογία 5 Κρόιτσμαν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 του υποφαινομένου υπέρ, κατά. Σας ευχαριστώ. Τροπολογία 12 Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται τροπολογία 19. Ζουβέν Αμπάντ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 των ιδίων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 11. Κρόιτσμαν ως προσθήκη. Υπέρ κατά, αποχές, επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 2, ε, συγγνώμη, τροπολογία 8, Κρόιτσμαν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική τροπολογία 2, από κάποιους συναδέλφους, ε, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα, πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 13, Κρόιτσμαν, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, ως προσθήκη ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 ως προσθήκη υπέρ, κατά, και αυτή εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 29 προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν 23 και περνάμε στην τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Και περνάμε στη συμβιβαστική 3. Ψήφι υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Άρα ολοκληρώνουμε με τις τροπολογίες και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Για τα πρακτικά έρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν 27 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια κύριε Κρότσμαν. So thank you all very much and I know... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω πως ο κύριος Κρότσμαν οπωσδήποτε θα υπερασπιστεί τις τροπολογίες μας στην Επιτροπή Βιομηχανίας για να συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Οπότε τελειώνουμε, τελειώσαμε τις ψηφοφορίες και είμαστε και νωρίς σε σχέση με το πρόγραμμά μας, οπότε θα διακόψουμε για λίγο οποίος ε, δεν θα μείνει για την έκθεση Μάιερ για το ε, δίκαιο των συμβάσεων και θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά. Uh, uh, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω πως όλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Σταν από την Κομισιόν που έχει εργαστεί πολλές φορές εδώ πέρα, ειδικά όσον αφορά την ε, καταναλωτική πίστη και χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε στον νέο ρόλο σας στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και βεβαίω είναι εδώ και ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάιερ που είναι ο εισηγητή μας για τη σημαντική αυτή γνωμοδότηση στην ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Και μετά από αρκετή συζήτηση καταλήξαμε σε μια συζήτηση ε, με βάση τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας ε, και νομίζω πως έχουμε κάποια αποκλειστική αρμοδιότητα στην απάντησή μας στο πράσινο βίβλο της Κομισιόν. Λείπουν οι σκιοδησηγητές, κυρία Στήλερ λείπει, κυρία Ρούλε είναι εδώ, χαίρομαι, κύριος Φόξ λείπει, αλλά θα πω εγώ κάποια λόγια, ξενοματώσω και ο κύριος Αλβίνη δεν είναι εδώ, οπότε... Όσον αφορά το συνολικό χρονοδιάγραμμα, όπως ξέρετε πρέπει να συμφωνήσει η διάσκεψη των Προέδρων για την συμφωνία που έχουμε κάνει εμείς με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αλλά δεν αναμένω δυσκολίες. Αυτό θα επιβεβαιωθεί, φαντάζομαι, στο Τρασβούργο της ερχόμενης εβδομάδας. Θα δώσω τώρα τον λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Μάιερ. Αν θέλετε να μιλήσει η Κομισιόν αμέσως μετά από εσά, νομίζω αυτό εξαρτάται από εσά. Άρα καλό είναι να ξεκινήσετε εσείς ως συζητητής είναι, το βρίσκεται σωστό, θέλετε να κάνετε μια εισαγωγή και μετά να ζητήσω τον κύριο εκπρόσωπο της Κομισιόν να κάνει μια εισαγωγή και να γίνει μια συζήτηση. Το δέχεστε αυτό και οι δύο. Ο κύριος Μάιερ λοιπόν και μετά ο κύριος Στάιν Okay, Mr. Meyer. Okay, Herr Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πράσινη βίβλος, δεν είναι λοιπόν άμεσο νομοθετικό ζήτημα αυτό το οποίο έχουμε. Μιλάμε για επιλογές που αντιμετωπίζουμε, τι θα μπορούσε να γίνει. Βλέπετε, πολύ υποθετικός λόγος. Συνολικά δεν είναι ευρύτατο έτσι, αυτή η πράσινη βίβλος, αλλά έχει πολύ εκρηκτικό υλικό. Όπως είπε και ο Μάλκομ, ο πρόεδρός μας, η αρμοδιότητα είναι από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εδώ και δέκα χρόνια τώρα στο πλαίσιο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ως μέλος ε, έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα, οπότε χαίρομαι που το συνεχίζω στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Συμφωνήσαμε πως ε, η αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς ισχύει για το σημείο 3.1 για τις συμβάσεις. Επίσης υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα για το 4.2.1, δηλαδή για το εάν το μέσο αυτό θα πρέπει να ισχύει και για συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και για συμβάσεις με καταναλώτες. Και επιπλέον μεικτή αρμοδιότητα στο 4.3 για το θέμα ποιος είναι, ε, ο, ποιο είναι το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του μέσου αυτού. Οπωσδήποτε όλοι έχουμε διαβάσει την Πράσινη Βίβλο. Έχετε δει λοιπόν ποια είναι τα θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε εδώ πέρα πάντα βεβαίω στο, πλάσιο, στο πλαίσιο της πράσινης αυτής βίβλου και όχι στο πλαίσιο κάποιας νομοθεσίας. Οπότε το ζήτημα είναι ποιος είναι ουσιαστικός τομέας εφαρμογής εδώ πέρα. Αν θα έχουμε μια στενή ερμηνεία, αν θέλουμε έναν ορισμό δηλαδή με βάση ένα ορισμό της σύμβασης εδώ πέρα. Για μένα είναι σαφές πως στην εσωτερική αγορά στις 27 ένομες τάξεις έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το πότε συνάπτεται μια σύμβαση. Οπότε λέει κάποιος ναι και το ναι αυτό είναι δεσμευτικό. Και βεβαίω το θέμα μετά είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε με τις ε, υποχρεώσεις, ε, τις συμβατικές ε, τα λοιπά την παροχή υπηρεσιών ή να σταματήσουμε αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς μετά ως βασικά συστατικά σημεία θα τα κάνουμε δεσμευτικά να μην είναι δηλαδή να αντικαθιστούν κάτι αλλά να είναι δεσμευτικά ως λύση για τα κράτη-μέλη ή θέλουμε να εφαρμόσουμε την επικουρικότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί ο καθένας να λέει ε, πως ε, είτε έχουμε εδώ πέρα μια σύμβαση είτε δεν έχουμε και αναλόγως να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Κατά την άποψή μου λοιπόν πρέπει να πάμε στην πλήρη εναρμόνιση και το θέμα είναι μετά ως ποιο βαθμό θα γίνει αυτό. Υπάρχει βεβαίω και η ερμηνεία η οποία διαφέρει σε πάρα πολλά σημεία, παραδείγματος χάρη όσον αφορά το τις συνέπειες, την ε, εξωσυμβατική ερμηνεία κτλ. Και μετά αν θα πρέπει να ισχύουν για συγκεκριμένα είδη συμβάσεων, π.χ. αγοράς, υπηρεσιών κτλ. ή αν θα πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής προς την κατεύθυνση ενός ε, ευρωπαϊκού αστικού κώδικα. Θεωρώ πως θα πρέπει να δούμε το τι είναι εφικτό άμεσα και το τι είναι πιο αναγκαίο να το κάνουμε και δεσμευτικό. Και βεβαίω αυτό το οποίο μετά εμπίπτει στην επικουρικότητα να ε, μην ε, το συμπεριλάβουμε σε τόσο δεσμευτικό χαρακτήρα. Για να βρούμε δηλαδή τη σωστή ισορροπία, το που χρειάζεται σαφήνεια προς όφελο του καταναλωτή και τη επιχείρησης βεβαίω, η οποία θα ξέρει τι προσφέρει και τι ε, δεσμεύεται εναντί του καταναλωτή. Και θα υπάρχουν βεβαίω και τα μέτρα προστασίας. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε το προτινόμενο πλαίσιο και όπως σας είπα, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα, ο χρόνος πιέζει, πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε τι θα είναι δεσμευτικό και τι θα αριθμιστεί στο πλαίσιο της επικουρικότητας. Τώρα οι λεπτομέρειες μετά, σε ποιο βαθμό θα τα ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα, ζητήματα μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά τα βασικά, τα θεμελιώδη ερωτήματα είναι νομίζω τα σημαντικότερα. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να εξηγήσει την πρότασή της, να μας πει πού δίνει εκείνη το βάρος και μετά να επανέλθω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, thank you very much for... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτή την ε, παρουσίαση. Και να δώσω το, λόγο στον κύριο Στάν Μαϊγερ ώστε να συνεχίσει με βάση τα όσα μας εξέθεσε ο κ. Μάιρ και να μας παρουσιάσει το ιστορικό και τις κεντρικές ιδέες που περιλαμβάνονται στο πράσινο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στη βάση αυτής της πράσινης βιβλίου πριν περάσω στις επιλογές που έχουμε. Γιατί η πράσινη βίβλος σαφώς δεν αποτελεί μια λύση που αναζητεί πρόβλημα, αλλά έχουμε διαπιστώσει αντιθέτως πάρα πολλά προβλήματα για τα οποία αναζητούμε συγκεκριμένες λύσεις. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με τις ε, συμβάσεις ε, των καταναλωτών, γιατί βρισκόμαστε βέβαια και σε αυτήν την επιτροπή και μετά θα πω και λίγα λόγια για τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στην πλευρά των επιχειρήσεων όσον αφορά τη Σύμβαση καταναλωτών για να αναφέρω ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πλευρά των επιχειρήσεων. Θέλω εδώ πέρα να τονίσω πως πρώτα απ' όλα δίνουμε βάρος στα πλεονεκτήματα για τις μικρές και τις μισές επιχειρήσεις που αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων και υπάρχει σαφής στατιστικός συσχετισμός μεταξύ της ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης ε, και του περιορισμού της ανεργίας και της πρόθεσης της καινοτομίας. Οπότε όταν μιλάμε και επικεντρωνόμαστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την οικονομία και μπορεί να συνεισφέρει ως ένα μικρό κομμάτι στη γενικότερη λύση για να βγούμε από την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τον Νοέμβριο είχε εγκριθεί τα νούμερα ανάπτυξης κομισιών και εκεί πέρα βλέπετε πως η μέση οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης ήταν 1,8%. Αν το συγκρίνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 2,7%, η Ιαπωνία 3,5%. Οι ΙΠΑ ήταν πολύ ισχυρότερες. Ε, και επηρεάστηκαν πάρα πολύ περισσότερο από την ε, κρίση, αλλά συνολικά είχαν μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ευρώπη. Και αν δούμε αυτό το 1,8% που είναι μέσος όρος, βλέπετε πως το, ε, όπως είπα, είναι μέσος όρος. Δηλαδή, είναι 1,8 γιατί κάποια κράτη-μέλη, όπως η Πολωνία, η Σουηδία, η Γερμανία, έχουν ανάπτυξη γύρω στο 4%. Δηλαδή, και το 1,8% το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα πολλά υποσχόμενο έγινε λόγω κάποιων μερικών κρατών που τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Αυτό όσον αφορά αυτή την πτυχή της Πράσινης Βίβλου και όπως σας είπα την, ε, το σκεπτικό που είναι να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα όμως συγκεκριμένα υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Όπως ξέρετε γιατί είναι ο τομέας αρμοδιότητάς σας, εάν βρεθούμε, παραδείγματο χάρη, στην θέση μιας μικρομεσαίας ε, επιχείρησης ε, η οποία θέλει ε, να πουλήσει κάτι συνοριακά, θα εφαρμόσει το δίκαιο της χώρας του αγοραστή και των δύο χωρών, όπως παραδείγματο χάρη αναφέρει το άρθρο 6 του κανονισμού Ρώμη 1, κάτι το οποίο βεβαίω είναι πάρα πολύ δύσκολο και κοστίζει γιατί θα πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνει ακριβώς η εκάστοτε εθνική νομοθεσία και βεβαίως θα πρέπει να μάθει η σύμβαση την οποία έχει ήδη έτοιμη, πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί για να είναι αφενός νόμιμη, για να ισχύει και στο άλλο δίκαιο, αλλά βεβαίως και πώς η σύμβαση αυτή θα είναι και οικονομικά συμφέρουσα για την επιχείρηση, γιατί βεβαίως ε, η γενική όροι με βάση του κάνει μια απόλυση μια επιχείρηση είναι βεβαίως νόμιμοι αλλά είναι και οι πιο συμφέροντες κάτι το οποίο βεβαίως δεν ταυτίζεται πάντα όταν απευθύνεται κανείς ε, και κινείται σε ένα άλλο νομικό πλαίσιο μιας άλλης χώρας. Στα τέλη του προηγούμενου έτους λοιπόν κάναμε μια έρευνα μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ρωτήσαμε Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια, τα 13 μεγαλύτερα εμπόδια για τις διασυνοριακές συναλλαγές και βλέπουμε πως τα πρώτα 10 εμπόδια τα οποία αναφέρθηκαν 6 από αυτά αφορούν το δίκαιο των συμβάσεων, το ενοχικό δίκαιο. Το πρώτο πρόβλημα βεβαίω ήταν πρώτα απ' όλα να διαπιστωθεί ποιο ήταν το εφαρμοστέο δίκαιο. 74% των ερωτηθέντων το ανέφεραν αυτό ως πρόβλημα. Μετά όμως, αμέσως μετά, ήταν η μετάφραση του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου με 68% και 65% τα έξοδα των δικηγόρων. Έλλειψη λοιπόν εμπιστοσύνης μετά στο ξενοδίκαιο, ο φόβος για δικαστικές περιπέτειες στην άλλη χώρα με ένα 58% και βεβαίως η δυσκολία διαπραγμάτευσης με τον αντισυμβαλόμενο και να συμφωνήσουν στο ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως όταν ρωτάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνεται σαφές πως τα εμπόδια του ενοχικού δικαίου είναι πάνω-πάνω στην λίστα των αιτιών που τις εμποδίζουν να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά τρεις στις τέσσερις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, δεν δραστηριοποιούνται διασυνοριακά για μια σειρά λόγων. Και κάποιους από αυτούς τους ανέφερα. Γνωρίζουμε όμως πως 50% αυτών των επιχειρήσεων θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν και θα το έκαναν εάν υπήρχε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ρωτήσαμε πιο λεπτομερώς όχι μόνο για ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και για τις επιλογές που αναφέρονται στην πράσινη βίβλο ρωτήσαμε παραδείγματο χάρη τις μικρομεσαίε αυτές επιχειρήσει. Ποιε επιλογές θα προτιμούσαν. Και ήταν σαφής η προτίμηση για ένα ευρωπαϊκό ενιαίο ενοχικό δίκαιο 88% όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνά μας μας είπαν πως θα προτιμούσαν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ενοχικό δίκαιο και αυτό το θεωρούν κάτι καλό ή πάρα πολύ καλό μάλιστα και 78% αυτών των επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούσαν ένα προαιρετικό μέσο πιθανότατα ή σχεδόν βέβαια εάν υπήρχε αυτό. αυτό αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο θέμα, το δεύτερο εμπόδιο, το δεύτερο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για όλες τις επιχειρήσεις συνολικά, είναι το θέμα της εκμετάλλευσης των διαφόρων πλέον εκτιμάτων της συνέργειας. Εάν υποθέσουμε πως ε, το προϊόν σας ε, ή την υπηρεσία σας ε, με κάποιον τρόπο ηλεκτρονικά. Πρέπει βεβαίως ε, να προσαρμόσετε τη σύμβαση. Εάν σκεφτείτε όμως πως με βάση μόνο ένα εθνικό, θα μπορούσατε να ε, κινήσετε με βάση μόνο ένα εθνικό δίκαιο και να έχετε μία μόνο ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα είχαμε φοβερές οικονομίες. Και μετά ρωτήσαμε πώς θα έβλεπαν αυτές τις οικονομίες, αυτές οι επιχειρήσεις και πάνω από το μισό των ερωτηθέντων μας είπαν πως βεβαίως θα είχαν τέτοιες οικονομίες, ε, γύρω στο 54% ε, σε διάφορους βαθμούς, τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει πως η πλειοψηφία των ε, ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όπως σας είπα αυτό δεν αφορά καν μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά όλες τις επιχειρήσεις συνολικά αν δει λοιπόν κανείς αυτά τα νούμερα, αντιλαμβανόμαστε πως πάνω από τις μισές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο όφελος οικονομικό από την εκμετάλλευση αυτών των συνεργειών. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά προβλήματα που ισχύουν ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έρχομαι τώρα στους καταναλωτές, που είναι νομίζω βασικό σημείο και της δικής επιτροπής. Στους καταναλωτές βλέπουμε πάλι δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι, και εδώ πέρα μπορώ να σας αναφέρω νούμερα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάναμε μια έρευνα και φτιάξαμε ένα καλάθι με 100 προϊόντα τα οποία αγοράζει συχνά ο καταναλωτή. Και είδαμε πόσα από αυτά τα 100 προϊόντα είναι διαθέσιμα στην εθνική αγορά online. Και θα ξεκινήσω με το πιο σοκαριστικό νούμερο. Στις μικρότερες εθνικές αγορές, Μάλτα και Κύπρο, 98 από τα 100 προϊόντα δεν ήταν διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην εσωτερική αγορά. Μπορεί να πει κανείς, εντάξει είναι δύο νησιά τώρα, είναι και μικρές αγορές, δεν αξίζει και τον κόπο. Σωστά αυτά. Αλλά αν δούμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αρχίζοντας να ανεβαίνει. Τα επόμενα 13 κράτη-μέλη μετά. Κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη αυτά τα 13 πάνω από τα 50 από τα 100 προϊόντα δεν ήταν πάλι διαθέσιμα και κάναμε έλεγχο μετά. Εάν πάει κάποιος σε άλλο κράτος μέλος, εξοικονομεί. Και είδαμε πως πάνω από το μισό αυτών των προϊόντων είχαν τουλάχιστον οικονομία τουλάχιστον, λέω, 10%. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει πως ο εκάστοτε καταναλωτής, ειδικά σε μικρές εθνικές αγορές, Πρώτον, έχει πολύ μικρή επιλογή. Δεύτερον, σε μη ανταγωνιστικέ τιμέ. Και τρίτον, πιθανότατα σε ελλειπή ποιότητα. Αυτό σημαίνει πως ο ανταγωνισμός, ειδικά για τα μικρά κράτη-μέλη, δεν λειτουργεί για τον καταναλωτή. Αγοράζουν και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά, δεν μπορούν να βρουν όλα τα προϊόντα τα οποία θα ήθελαν. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι πως κάναμε, ε, ψωνίσαμε ανώνυμα και προσπαθήσαμε να κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές, γύρω στις 11.000 συναλλαγές. Και γύρω στο 61% των συναλλαγών δεν έγιναν, δεν εκτελέστηκαν. Και για ποιο λόγο, βεβαίως υπήρχε μια σειρά λόγων, αλλά σημαντικό κομμάτι ήταν πως υπήρχε άρνηση να πουλήσουν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Φανταστείτε πως είστε, ξέρω εγώ, καταναλωτής Λετωνία, ας πούμε. Είστε Λετωνός καταναλωτής και θέλετε να αγοράσετε κάτι στο ίντερνετ από ένα πολωνικό γερμανικό site, μια μικρο... μεσαία επιχείρηση. Πάτε στο site, βρίσκετε το προϊόν, το βάζετε στο καλάθι και κάποια στιγμή βλέπετε στην οθόνη ε, να συμπληρώσετε τα δεδομένα σας. Πού μένετε, πώς θα πληρώσετε, πού παραδίδονται κουτουλού. Πατάτε λετωνία, τσακ, αλλάζει η οθόνη και λένε «Α, δεν πουλάμε στη Λετωνία». Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν έχει νόημα, εννοώ δεν συμφέρει για πολλές επιχειρήσεις να στείλουν τα προϊόντα σε άλλες εθνικές μικρομεσαίες αγορές, γιατί για τους λόγους που ανέφερα. Οπότε αυτά είναι τα προβλήματα που ήθελα να αναφέρω. Τώρα δεν θέλω να επιμείνω πάρα πολύ ε, να μπω πάρα πολύ στην ε, πράσινη βίβλο. Έχουμε κάποιες επιλογές, 7 επιλογές που νομίζω πως καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πιθανών λύσεων. Έχουμε από μια μακροσκελέστατη, θα έλεγα, ε, διαβούλευση. Τόσα χρόνια που δουλεύω στην Κομισιόν δεν έχω δει 7 μήνες περίοδο διαβούλευσης για να φροντίσουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να το συζητήσουν, να πούν την άποψή τους, να ακουστούν. Κάποια α, πραγματάκια να πω για μία επιλογή, γιατί αυτή τη στιγμή ακούω πάντα τα ίδια ερωτήματα. Δηλαδή, αυτό το προαιρετικό μέσο, εάν θα είναι δηλαδή ε, μια σύσταση. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί αυτό. Και εδώ πέρα έκανε μια ακρόαση η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όπου συζητήθηκαν όλα αυτά. Οπότε να σας πω πώς θα λειτουργήσει αυτό το θέμα. Το σκεπτικό είναι το εξής. Να ξεκινήσουμε από τις σκέψεις ε, που είχαμε για αυτά τα προβλήματα και να διαθέσουμε ένα μέσο το οποίο δεν θα εναρμονίζει, δεν θα υποκαθιστά το εθνικό δίκαιο και δεν θα επιβάλλεται εάν δεν το θέλουν τα συμβαλώμενα μέρη. Οπότε θα... δεν θα έχει άρα κόστος για εκείνους οι οποίοι δεν το επιθυμούν, αλλά μόνο για εκείνους οι οποίοι θα το επιλέξουν ως εφαρμοστέο δίκαιο για την σύμβαση την οποία θα συνάψουν. Και θα το επιλέξουν αυτό και θα το κάνουν μόνο εάν έχουν ένα οικονομικό πλεονέκτημα. Κλασική δηλαδή περίπτωση win-win, αμοιβαία εποφελής. Θα το επιλέξουν δηλαδή τα μέρη μόνο εάν είναι και τα δύο πεπισμένοι πως έχουν όλοι οικονομικά πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα, βεβαίω για την επιχείρηση ότι γλιτώνουν κόστος, αυτό το οποίο ανέφερα πριν, ανέφερα τα προβλήματα και για τον καταναλωτή υπάρχει αφενός το οικονομικό όφελος το οποίο ανέφερα, αλλά και νομικά πλεονεκτήματα, γιατί βεβαίως, βεβαίως και ο καταναλωτής θα το επιλέξει μόνο αν έχει πραγματικά πλεονεκτήματα. Και όχι μόνο οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά και νομικά πλεονεκτήματα. Και ποια θα είναι αυτά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πως έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και όχι μόνο υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή με την έννοια τη συνήθη. Αυτό το οποίο λέμε συνήθω και είναι φίλο ψυχής, αλλά ουσιαστικό. Δηλαδή ένα επίπεδο το οποίο θα βελτιώνει την κατάσταση του καταναλωτή σε σχέση με το υφιστάμενο και εκτιμένο και την εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν θα είναι πραγματική βελτίωση για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Επιπλέον πρέπει να προσέξουμε το εξή. Να δούμε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό γιατί οι καταναλωτές λένε πως το θέμα είναι και πώς εφαρμόζεται το δίκαιο αυτό στην πράξη και το δικαίωμα το οποίο έχω και η Κομισιόν είδε πως το τέταρτο τρίμηνο αυτού του έτου σκοπεύει να καταθέσει ένα μέσο για τις, α, τους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς για να υπάρχει δηλαδή μια σύνδεση μεταξύ ενός α, τέτοιου προαιρετικού μέσου και ενός απλού φτηνού τρόπου μέσου εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Και τέλος, ψηφιακά δικαιώματα. Συζητήσατε ήδη πριν γι' αυτό και εδώ πέρα πράγματι έχουμε μια δυνατότητα να πούμε πως αυτά τα δικαιώματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και τα οποία πόσο ξέρουμε δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα επαρκώς στα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα ευρωπαϊκό μέσο του ε, ενοχικού δικαίου που δεν υπάρχει ούτε στο κεκτημένο ούτε στο εθνικό δίκαιο να υπάρχει δυνατότητα για τον καταναλωτή να το επιλέξει. Οπότε για τους καταναλωτές δεν υπάρχουν όπως είπα οικονομικά μόνο ωφέλη που θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να αγοράσει κάποια προϊόντα παραπάνω σε καλύτερη τιμή, αλλά και ουσιαστική νομική προστασία. Και θα ήθελα να κλείσω εδώ πέρα, ε, να πω μόνο δύο προτάσεις για τις ε, συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Ξέρουμε πως τα προβλήματα τα οποία ανέφερα ε, ισχύουν κυρίως για τις συμβάσεις λιανικής. Μεταξύ επιχειρήσεων είναι λιγότερα τα προβλήματα, γιατί βεβαίως εκεί πέρα υπάρχει η δυνατότητα ελευθερίας των συμβάσεων και μπορούν να επιλέξουν τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις. Σε τι οδηγεί αυτό. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά στο ότι η ισχυρότερη πλευρά από τις δύο ορίζει το εθνικό της δίκαιο ως το δίκαιο το εφαρμοστέο σε αυτή τη σύμβαση. Θέλει να κάνει κάτι κομισιόν εδώ πέρα. Όχι. Γιατί, γιατί το ρυθμίζει η αγορά και αυτό είναι κάτι το θετικό, αλλά βρεθείτε λίγο στη θέση της επιχείρησης η οποία είναι ασθενέστερη εδώ πέρα. Και εδώ πέρα πάντα, ε, κατά κανόνα εν πάση είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρομεσαία αυτή επιχείρηση πρώτα απ' όλα θα έχει όλα αυτά το κόστος το οποίο προανέφερα και μια κάποια δυσπιστία. Γιατί η άλλη μεγαλύτερη επιχείρηση επέλεξε το δικό της δίκαιο και διαμόρφωσε ανάλογα τη σύμβαση έτσι ώστε να είναι οι συμφερότεροι για εκείνην. Εάν τώρα αυτές τις δύο επιχειρήσεις ε, έχουν στη διάθεσή τους ένα ουδέτερο, εάν θέλετε, δίκαιο, έχουμε ένα εμπόδιο το οποίο φεύγει. Γιατί όπως σας είπα, 55% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είπαν πως είναι ακριβώς πρόβλημα η διαπραγμάτευση όσον αφορά το εφαρμοστείο δίκαιο και υπάρχει αυτή η δυσπιστία και βέβαια αν δεν θέλει κάτι τέτοιο η μεγάλη επιχείρηση, τότε θα έχουμε ούτως ή άλλως πλεονέκτημα στην περίπτωση στην οποία τι συμβαίνει και οι δύο πλευρές είναι μικρές ή μικρομεσαίε. μικρομεσαίες. Ας φανταστούμε, ξέρω εγώ, μια γαλλική επιχείρηση από την Αλσατία που πουλάει στην άλλη μεριά του Ρήνου στη Βάδη Βερτεμβέργη. Δύο μικρές επιχειρήσεις και καμία δεν είναι ισχυρότερη από τις άλλες. Αυτές οι δύο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα το οποίο όπως σας είπα ανέφεραν 55% των επιχειρήσεων τις οποίες ερωτήσαμε, να το αποφύγουν και να διαλέξουν ένα ουδέτερο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτά είναι τα προβλήματα λοιπόν τα οποία διαπιστώσαμε, αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες προτείναμε και βεβαίως αυτή είναι η διαβούλευση η οποία έχει γίνει. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ χρήσιμη εισαγωγή σας. Δύο πράγματα πριν ξεκινήσω τη συζήτηση θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τα στατιστικά στοιχεία που μας δώσετε ήταν πολύ ενδιαφέροντα από το Ευρωβαρόμετρο που έρχονταν. Έχετε στοιχεία από κάποιες έρευνες, έτσι. Είναι κάποια στοιχεία από μια ξεχωριστή έρευνα, τα έχετε δημοσιεύσει κάπου, θα μπορούσαμε να τα προμηθευτούμε γιατί είναι χρήσιμα. Και δεύτερον, Μιλήσατε για μια πιο ευρεία μελέτη επιπτώσεων. Σε σχέση με τις προτάσεις αυτές, ε, συμπληρωματική θα είναι αυτή ίσως. Ε, θα ήθελα να μας πείτε και για αυτά αργότερα, θα σας ξαναδώσω το λόγο. Είναι έτσι πρακτικά θέματα που μας ενδιαφέρουν, αλλά ας ε, ξεκινήσουμε ένα γύρο σχολείων από τους συναδέλφους κύριος Μάγερ έκανε την εισαγωγή του, σκιώδης για τους πρασίνους είναι η κυρία Ρούλε νομίζω. Ο κύριος Σμιτ δεν είναι εδώ, Στάιλερ επίσης δεν είναι εδώ. Άρα, κυρία Ρούλε, ο σκιώδης ηγέτρια από τους πρασίνους θα έχετε το λόγο και εγώ θα μιλήσω επίσης κασότασε και εγώ τον κύριο Φόξ. Και κάποιοι άλλοι ομιλητές, Μάντες Κρόιτσμαν, κάποιος άλλος και φυσικά και ο Μάγερ ε, θα δευτερολογήσει. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Ρούλη όμως. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μάιερ, γιατί τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Και νομίζω πως σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, δηλαδή να δούμε πού υπάρχει ε, ανάγκη να δράσουμε επιγόντως. Εγώ θεωρώ πως υπάρχει ένας κίνδυνος ε, με την ευρύτερη προσέγγιση της ε, Κομισιόν να καταλήξουμε ε, σε μία ανάλογη κατάσταση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σβάμπ. Δηλαδή να συζητάμε, να συζητάμε και τελικά να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε παρά ελάχιστα. Μιλήσατε για μια κατάσταση ε, αμοιβαία υποφελία, αλλά δεν θα μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν όλοι. Το θέμα είναι ποιο θα την κερδίσει. Είπατε πως βεβαίως πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή έτσι ώστε οι καταναλωτές να δεχτούν να συμμετάσχουν. Αλλά βεβαίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν μόνο εάν δεν ανέβει το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Αυτά τα ζητήματα τα, συζητήσαμε με τον κύριο Σφάμπ και φοβάμαι πως ξανά επαναλαμβάνεται η ίδια συζήτηση. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πράγματι ποια είναι αυτά τα αναγκαία και κατεπήγοντα ζητήματα που θέλουμε να ρυθμίσουμε. Αυτή την προσέγγιση θα ήθελα εγώ να ακολουθήσει η Επιτροπή. Θα μιλήσω κι εγώ αυτή τη στιγμή εξ ονόματος της μου. Θέλω να πω ότι συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που μόλις είπε η κυρία Ρούλε. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εδώ για να μην ξεκινήσουμε μια πολύ μακρά επιχειρηματολογία πάλι για μια πρόταση εναρμόνισης. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν επενδυθεί πόροι και οικονομικοί αλλά και εμπειρογνωμοσύνης. Και εγώ όταν πρωτοήλθα εδώ το 99 πάλι συζητήτω το θέμα αυτό και νομίζω ότι ένα από τα θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι μπορεί να περάσουμε σε κάποιες κοινέ αρχές, αλλά τα νομικά συστήματα και η εφαρμογή, εκείνο το πρόβλημα στα κρατημέλη, είναι διαφορετική. Και αυτό μας δυσκολεύει και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το να υπάρχουν λοιπόν εργαλεία αυτή προσέγγιση της εργαλειοθήκης. Νομίζω ότι μας δίνει δυνατότητα, τη δυνατότητα να ελέγξουμε στην πράξη κάποιες έννοιες, να δούμε πόσο πολύτιμες μπορεί να είναι. Και μπορούμε και να κάνουμε έτσι παρατηρήσεις για κάποια περίοδο και μετά να ξεκινήσουμε κάτι πιο φιλόδοξο. Το έγγραφο, όπως το βλέπω, γενικά νομίζω ότι εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στο καταναλωτικό δίκτυο στην νομοθεσία για τους, για, για, τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τις βάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, λέει το κείμενο ότι ήδη οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν κάποια τυποποιημένα μέσα ε, στο πλαίσιο των ισχυουσών συμβάσεων και ίσως το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο θα ήταν κάτι επιπλέον, κάτι συμπληρωματικό. Ίσως λοιπόν και πάλι να εστιάσουμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν στους καταναλωτές και γνωρίζουμε ποιε είναι οι δυσκολίες, τις αντιμετωπίζουμε ήδη. Έχουμε την ε, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Έχουμε την οδηγία για την καταναλωτική πίστη, ο κύριο Στάντερμαϊρ και κάποιοι άλλοι. Είμαστε βετεράνοι για αυτή, σε αυτή τη διαδικασία που κρατάει πολύ καιρό. Δεν ξέρω, μπορεί να πείτε ότι είναι βρετανική η προσέγγιση, ότι πρέπει να είμαστε πιο πραγματιστές, πιο ρεαλιστές, αλλά καλό θα ήταν να βγάλουμε από το εργαστήριο αυτές τις ιδέες και να τις δοκιμάσουμε στην πράξη, για να δούμε τι αξίζουν τελικά. Εγώ προσωπικά, και όχι μόνο εγώ, αλλά και η ομάδα μου, δεν είμαστε υπέρ, αντιθέτω είμαστε κατά της τρίτης επιλογής ε, που προτείνει η Κομισιόν. Ίσως η καλύτερη λύση θα ήταν κάποια κάποιο συνδυασμό των πρώτων δύο επιλογών. σε επιλογή 1 και 2. Σίγουρα θέλουμε να γίνει μια πιο συνεκτική ανάλυση του κόστους, ε, των επιπτώσεων που συνεπάγονται όλα αυτά. Και από την άλλη νομίζω ότι ως έχει η πρόταση αυτή τη στιγμή, έχει αναπτυχθεί, θα έλεγα, υπό εργαστηριακές συνθήκες ε, και δεν έχει εκτεθεί σε κάποιες πρακτικές πραγματικότητες που έχουν να κάνουν δηλαδή με το πώς δουλεύει μια πολύπλοκη αγορά. Και καλό θα ήταν να έχουμε μια πιο διευρυμένη θα έλεγα διαδικασία ανάπτυξης. Δεν θέλω να υψέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά να θα συνεργαστούμε με τα χάρας με τον κύριο Μάγερ και στη συνέχεια. Επόμενος είναι ο κύριος Σβάπ και μετά Μέντες και Κρόιτς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ βεβαίως με αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι και εσείς βεβαίως, αλλά θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα πως η ανάλυση των προβλημάτων που έκανε η Κομισιόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των καταναλωτών από τις μικρές χώρες με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Και ο καθηγητής Μόντι κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα στην έκθεσή του η οποία νομίζω υποστηρίχθηκε σε όλα τις τα ουσιαστικά σημεία από την Επιτροπή μας. Οπότε, όσον αφορά τους στόχους, το βασικό είναι εάν μπορούμε να εφαρμόσουμε πραγματικά και αν έχουμε όντως τους ίδιους στόχους και τα ίδια μέσα. Οπότε το ερώτημά μου προς τον κύριο Στάινμαϊερ είναι πώς θα μπορέσει η Κομισιόν να σχηματίσει εκείνες τις πολιτικές πλειοψηφίες που υπήρχαν για την ε, οδηγία δικαιωμάτων των καναλτών. Γιατί τα ε, σημεία εκεί πέρα ήταν πως είπανε τότε πως δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο αύξηση τόσο των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι έχει αλλάξει ως προς αυτό. Δεύτερον, τι προσθέτει ως πρακτική προσθέμενη αξία αυτή η πρόταση. Με τα δικαιώματα των καναλτών. Πάντα η, ήταν οι σύνδεσμοι των επιχειρήσεων, π.χ. η ΓΕΣΕΒΕ, η αντίστοιχη στη Γερμανία κτλ. Πάντα έκαναν μία πρόταση. Και έλεγαν μην τα κάνετε και πολύ... Έτσι πάντα ήταν περιορισμένες οι φιλοδοξίες τους. Τώρα για τα νομικά επιχειρήματα, νομίζω πως αυτά είναι υπέρ της πλήρους εναρμόνισης, αλλά βλέπουμε πως δυστυχώς προς τα εκεί δεν πάει κανείς παρά τα όσα επιθυμούσε η Κομισιόν. Και υπάρχει νομίζω και μια σαφής, ξεκάθαρη νομική βάση. Και τέταρτον, για τον τομέα της εφαρμογής. Νομίζω πως και οι ενώσει των καταναλωτών στο τέλος θα εξετάσουν ποιο δίκαιο είναι το ε, συμφερότερο και θα επιλέξουν είτε το εθνικό είτε το ε, προαιρετικό μέσο όπως είπατε. Δεν ξέρω εάν αυτή είναι η κατάσταση την οποία θέλαμε. Οπότε με την ανάλυση συμφωνώ οπωσδήποτε. Το θέμα είναι εάν ε, οι λύσεις είναι αυτές οι οποίες προτείνετε. Ευχαριστώ. Κύριος Μάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ φυσικά με πολλούς από τους ομιλητές και πρέπει να σας πω ότι αυτά που είπε ο εκπρόσωπος Επιτροπής, κάποια από αυτά με εξέπληξαν διότι και με χαροποίησαν που τα άκουσα γιατί εδώ και χρόνια τα λέμε στην Επιτροπή μας. Όταν όμως πρέπει να συζητήσουμε πραγματικά ε, οδηγίες ή κατά προτίμηση κανονισμούς, όλοι τότε επικεντρωνόμαστε στην εθνική προσέγγιση και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κατά την άποψή μου λοιπόν, ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι η τέταρτη επιλογή. Δηλαδή, δύο προσεγγίσεις, πρώτα εθνική προσέγγιση και μετά μικρομεσαίες και καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά, κανονισμό, προαιρετικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως οι καταναλωτές σήμερα δεν εμπιστεύονται ε, τις δεσνοριακές αγορές γιατί δεν ξέρουν ε, τι μπορούν να αναμένουν ούτε από το νομικό σύστημα ούτε από τα προϊόντα που θα τους ε, σταλούν. είναι το πρόβλημα. Είναι ένα θέμα που το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό και για την χρονομίσθωση και τώρα βλέπουμε ότι κάθε κράτος μέλος έχει κάνει τα δικά του σε εθνικό επίπεδο, άρα δεν υπάρχει εναρμόνιση ουσιαστικά. Ουσιαστικά δηλαδή παρακάμπτεται ο ορισμός και τελικά στο μέλλον έχουμε κανονισμούς που δεν εφαρμόζονται. Γιατί δεν το θέλει το Συμβούλιο, δεν το θέλουν και αρκετοί συνάδελφοι αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη, ένα τρόπο σκέψης και μια νέα αγορά, μία μόνο προσέγγιση είναι αυτή που θα λειτουργήσει, δηλαδή κανονισμός. σε ευχαριστώ. Εσείς πράγματι είσαστε συνεπέστατος ε, στην ε, άποψή σας. Ο κύριος Κρόιτσφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο κύριο Σβάμπ. Η ανάλυση είναι ξεκάθαρη, αλλά η λύση, ε, για αυτήν έχω αμφιβολίες εάν μιλήσετε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν θέλετε να τις προσελκύσετε με ένα απλό καθώς πράγματι ναι, πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια, αλλά αν από την άλλη θέλετε να αυξήσετε την προστασία του καταναλωτή, δεν θα ε, προσελκυστούν γιατί βεβαίως ζυγίζουν το όφελος και τον κίνδυνο και αν ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αφήνουν την ευκαιρία κατά μέρος να περάσει. Πρέπει να σκεφτείτε πως οι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις δεν έχουν πρόβλημα, έχουν θυγατρικές, ξέρουν τις δομές επιτόπου ή έχουν εξαιρετικούς δικηγόρους. Αλλά και αυτές ακόμα ζυγίζουν ποιες είναι οι ευκαιρίες και κινούνται αναλόγως. Αλλά μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα διατρέξει τον κίνδυνο του υψηλότερου αυτού επίπεδου προστασίας του καταναλωτού ή των ομαδικών αγωγών. Όπως ξέρετε και στη Γερμανία πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ήταν... Θα ήταν ηρωνικό να πάμε προς τα, προς τα εκεί. Οπότε είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μάιρε. Όλοι συμφωνούμε, θέλουμε να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά και αν τα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση που θα βοηθήσει τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις, θα τις προσελκύσει να κάνουν περισσότερες προσφορές σε άλλα κράτη-μέλη μέσω του διαδικτύου ή δεν ξέρω πώς. Οπωσδήποτε θα είναι θετικό αυτό και για τις επιχειρήσεις αυτές και για τον καταναλωτή. Αλλά φοβάμαι πως δεν θα γίνει τίποτα γιατί διαπιστώσαμε με τις έρευνες πως ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το ίντερνετ και τα λοιπά σύγχρονα μέσα πολύ επιφυλακτικά και όχι όπως ε, θα φανταζόμασταν. Ευχαριστώ κάποιος άλλος. Ίσως να, δώσω ξανά το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και μετά ο κύριος Μάγερ ε, θα συνοψίσει και θα μας μιλήσει για τα επόμενα βήματα και για το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να σας ευχαριστήσω και για τα ευγενικά σας ε, λόγια στην αρχή και για την οδηγία που είπατε κι εσείς για τους καταναλωτές και θα τη χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να πω κάτι που θέλω. Σε ό,τι αφορά όμως ε, κύριε Πρόεδρε τα πρώτα τρία σημεία που θίξατε από πού ε, Έχουμε τα στοιχεία. Εσείς μιλήσατε για έρευνα, ε, για τη μελέτη επιπτώσεων και για το ευρωβαρόμετρο. Λοιπόν, πριν υποβάλουμε την πράσινη βίβλο είχαμε κάποια προκαταρκτικά στοιχεία, αλλά βέβαια για να κάνουμε τη μελέτη επιπτώσεων να δρομολογήσαμε διάφορες έρευνες, ε, τέσσερις ε, βασικά έρευνες, δύο ευρωβαρόμετρα ήταν αυτά και επίσης μία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μία γενικά για τις επιχειρήσεις. Τέσσερις λοιπόν έρευνες. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στη θέση μας, ακόμη. Όταν θα τα συγκεντρώσουμε όλα, θα τα δημοσιεύσουμε. Τα λάβαμε όλα τα Χριστούγεννα και επομένως μέσα στο μήνα θα τα έχετε, ε, θα τα δώσουμε στην ε, γραμματεία σας μέσω μια σύνδεσης γιατί εμείς θα τα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο. Βέβαια θα έχουμε και άλλα δεδομένα. Αυτό το μήνα θα έχουμε περισσότερα δεδομένα και βέβαια θα τα δημοσιεύουμε όταν θα τα λαμβάνουμε στην ιστοσελίδα μας. Έτσι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Και βέβαια θα τα χρησιμοποιήσουμε για τη μελέτη μελέτης, ε, για την μελέτη επιπτώσεων. Ξέρουμε ότι είναι πολύπλοκο το σχέδιο για τη μελέτη επιπτώσεων ξέρουμε ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να αναλύσει τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις σε βάθος. Ήδη ξεκινήσαμε να εκπονούμε τη μελέτη επιπτώσεων και θα συνεχιστεί το έργο αυτό και φέτος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ήδη ε, ξεκινήσει. Τώρα περάσω στα γερμανικά. Για να απαντήσω σε κάποια από τα άλλα ερωτήματα. Δεν θα τα πάρω με χρονολογική σειρά. Θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω. Πρώτα απ' όλα για αυτό το οποίο είπε η κυρία Ρούλε και ο κύριος Κρόιτσμαν ανέφεραν και οι δύο πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν έχουν ένα μέσο απέναντί τους που προσφέρει υψηλότερη προστασία του καταναλωτή, δεν θα το επιλέξουν. Γιατί λέτε πως αυτό σημαίνει κίνδυνο ή κόστος, κύριε Κρότσμαν. Εν μέρη συμφωνώ, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Εν μέρη έχετε δίκιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται πάντα, σγίζουν δύο πράγματα. Δηλαδή αφενός είναι πολιτές έναντι του καταναλωτή, από την άλλη είναι αγοραστές σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι εταίροι. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό και από τις δύο πλευρές. Και ε, βλέπουμε πως στη συζήτηση έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Μερικές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κατά της υψηλότερης προστασίας των καταναλωτών, αλλά μιλάμε για διατάξεις που θα τις βοηθήσουν, παραδείγματος χάρη για περισσότερες Πληροφορίε σε σχέση με τι μεγαλύτερε επιχειρήσει τότε είναι υπέρ. Οπότε αυτή είναι η θέση στην οποία βρίσκονται οι μικρόμισε επιχειρήσει Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό συμφωνώ μαζί σα πω πράγματι ε, πως ε, αν τις δούμε ε, ως πολιτές πράγματι αυξάνεται το κόστος. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για την επιλογή αλλά πρέπει να δούμε το προαιρετικό αυτό μέσο, γιατί δεν εξαναγκάζουμε καμία μικρομεσαία επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το προαιρετικό μέσο. Είναι κάτι το οποίο θα ζυγίσουν. Θα δουν αφενός τα πλεονεκτήματα, τη νομική ασφάλεια, τη μείωση του κόστους και από την άλλη πιθανώς το ε, υψηλότερο επίπεδο που του καταναλωτή σε σχέση με το εθνικό του Θα διαλέξουν και θα επιλέξουν το συμφερότερο. Αλλά, και εδώ πέρα είναι η ουσιαστική διαφορά και έρχομαι στον κύριο Σφαμπ, αυτή είναι η βασική διαφορά έναντι της πλήρους εναρμόνισης. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά λοιπόν για το γιατί θα μπορούσε να είναι ευκολότερο να έχουμε ένα τέτοιο προαιρετικό μέσο, γιατί, γιατί οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές τελικά αποφασίζουν εάν θα δεχτούν αυτό το κόστος, γιατί από την άλλη σε αντιστάθμισμα θα λάβουν κάποια άλλα πράγματα, μεγαλύτερη προστασία, καλύτερες τιμές κτλ. Η διαφορά δηλαδή με την εναρμόνιση είναι πως δεν το επιβάλλουμε σε όλες τις επιχειρήσεις, ακόμα και αυτές που δεν το θέλουν, αλλά μόνο αυτοί οι οποίοι το θέλουν θα υπομισθούν το κόστος και διαλέγουν αξίζει τον κόπο και το κόστος και έτσι νομίζω μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, να διαλέξουν οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Θέλουμε δηλαδή να τα αφήσουμε στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να διαλέξουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ένα μέσο το οποίο πιθανώς θα προσφέρει οικονομικά πλεονεκτήματα. Για να έρθω τώρα στο δεύτερο σημείο του κυρίου Σβάμπ για τις πολιτικές πλειοψηφίες. Και εδώ πέρα μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε μία μικρή προσωπική παρέκβαση. Εγώ διαπραγματεύθηκα την ε, Οδηγία Προσφυσίας των του 1999 στο Συμβούλιο και ήταν ελάχιστη εναρμόνιση και η καταναλωτική πίστη τη σχετική οδηγία που ήταν η πρώτη οδηγία η οποία είχε πλήρη εναρμόνιση όσον αφορά το ενεργικό δίκαιο. Και ήταν σαφώς δυσκολότερη, όπως ξέρετε, να εγκρίνουμε την οδηγία περί καταναλωτικής πίστης. Γιατί επρόκειτο περί πλήρους Και στο Συμβούλιο όλα τα κρατη είπανε π.χ. στον ε, κατάλογο των ε, πληροφοριών θέλουμε αυτό και το χύψη και το τάδε γιατί ήταν ε, στην εθνική μας νομοθεσία. Υπήρχε ακριβώς αυτή η διάθεση να βάλει ο καθένας τα πάντα γιατί επρόκειτο περί εναρμόνισης και ξέραν όλα τα κρατη πώς θα αλλάξουμε το δίκαιό μας και κάθε υπουργός που πήγαινε πίσω στη χώρα του έπρεπε να πει στα επιμελητήριά του, είτε ήταν επιμελητήρια είτε ήταν καταναλωτές, γιατί συμφωνήσαμε στο χύψη πράγμα. Με το προαιρετικό μέσο είναι αλλιώς τα πράγματα. Με το προαιρετικό μέσο δεν αλλάζει το εθνικό δίκαιο. Ξακολουθεί να υπάρχει, μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται και επιχειρήσεις που δεν θέλουν να το εφαρμόσουν δεν έχουν κόστος. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και από πολιτική σκοπιά νομίζω θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πλειοψηφίε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε. Αλλά νομίζω αυτή είναι η βασική διαφορά με την πλήρη εναρμόνιση. Και τώρα να αναφερθώ σε κάτι άλλο το οποίο είπε ο κύριος Σβάμπ για το ότι οι ενώσει θα εξετάσουν ποιο μέσο είναι το καλύτερο. Οπωσδήποτε, ναι, και ε, έτσι πρέπει να είναι. Δεν λέει κανείς τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να εκπληρώνουν τον θεμητό και θεσμικό τους ρόλο. Και μετά ο καταναλωτής και η επιχείρηση βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ συγκεκριμένης κατάστασης. Θα αγοράσω αυτό το προϊόν που μου προσφέρεται από ένα άλλο κράτος μέλος εάν δεν το βρίσκω στη χώρα μου. Έτσι. Εάν είναι π.χ. 10% φθηνότερο και εάν έχω ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ίσως και υψηλότερο από το εθνικό μου επίπεδο. Και ίσως να είναι κάπως χαμηλότερο από κάποια κορυφαία κράτη. Γιατί, αυτή θα γίνει μετά. Θα υπάρχει η δυνατότητα τα συμβαλόμενα μέρη να το αποφασίσουν αυτό. Ο καταναλωτής και ο έμπορος. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Και τι συμβαίνει? Τίποτα. Δεν έχουν κόστος. Μπορούν να συνεχίσουν να απολούν και να αγοράζουν με βάση το εθνικό τους δίκαιο και η κατάσταση είναι αυτή η οποία ήταν πριν. Δηλαδή δεν τους αφαιρούμε τίποτα, τους δίνουμε μια επιπρόσθετη δυνατότητα που προστίθεται στο εθνικό δίκαιο. Και νομίζω πως και οι ενώσεις των επιχειρήσεων θα πούνε στα μέλη τους δείτε αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει. Και θα κάνουν αυτή την ανάλυση και θα πούνε σχέση με το εθνικό μας δίκαιο, το προαιρετικό μέσο εδώ είναι υψηλότερο, εκεί είναι χαμηλότερο και λάβετε την απόφασή σας. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν. Να μην πρώτα απ' όλα εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Αυτό είναι σαφώς. Πρέπει να υπάρχει μια υψηλή εγγύηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών καταναλωτών υψηλότερη προστασία από αυτή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως πράγματι κύριε Κρότσμαν αυτό μπορεί να είναι κόστος για την επιχείρηση αλλά μπορεί η επιχείρηση να το ζυγίσει, να πει τι θα μου προσφέρει και τι με συμφέρει εμένα. Να πουλήσω και ε, να είναι πιθανώ ακριβότερο με την ψηλότερη προσοχή του καταναλωτή ή με συμφέρει πράγματι να απευθυνθώ στου πάντε με μία πλατφόρμα πληροφορική. Ευχαριστώ. Πολύ, πολύ ωραία μα τα είπατε κύριε Στάινμάγερ. Ε, πολύ καλά κάνετε τη δουλειά πολιτή εδώ για αυτό το εργαλείο, το μέσο. δεν είμαστε πλήρω της πλήρως εναρμονισμένης πρότασης. Μιλήσαμε για την ε, μέγιστη δυνατή εναρμόνιση. Τέτοια κατεύθυνση έχουμε ακολουθήσει και με την οδηγία δικαιωμάτων του καταναλωτή. Επτά χρόνια μας πήρε για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Ανησυχία για μας ε, όλους είναι ότι ακόμα και η συμφωνία για ένα προαιρετικό ε, μέσο μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Γι' αυτό και εγώ τώρα προσπαθώ να σα πουλήσω τη δική μου ιδέα, ότι ίσω θα πρέπει να κάνουμε κάποια δουλειά ανάπτυξη. δηλαδή να έχουμε πρώτα ένα, μια εργαλειοθήκη και μετά αυτό θα παίξει το ρόλο πρόδρομου στο μέσο. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι θα πρέπει να βουτήξουμε με τα μούτρα σε κάτι τέτοιο. Αλλά ποιος ξέρει. Η Επιτροπή θα αποφασίσει τελικά. Και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον Hans Πίτερ Μάιερ για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους που έλαβαν το λόγο. Γιατί βεβαίως ο καθένας έχει δίκιο από τη σκοπιά του. Αλλά θα θέλαμε να συνοψίσουμε όσον αφορά τους καταναλωτές. Μικρή επιλογή, πολύ ακριβά τα πράγματα. Αυτή είναι η βασική λόγη. Και λέει κάποιος πως δεν, πολλά, δεν πουλάω π.χ. στη Λετωνία και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Όλα αυτά είναι σωστά. Και ένα προαιρετικό μέσο είναι επίσης μια καλή ιδέα επί της αρχής. Και βέβαια το ερώτημα είναι το τι θέλουμε αλλά τι θα γίνει στην πράξη εάν γράψει κάποιος πως αυτό το δίκαιο ισχύει και αν θέλει ε, το δέχεται ο καταναλωτής και ε, αλλιώς δεν έχει καμία επιλογή. Οπότε το θέμα είναι τι θέλουμε να έχουμε εδώ πέρα στην πράξη. Εάν θέλουμε να δώσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα στον καταναλωτή, τι χρειαζόμαστε ένα νέο αστικό κώδικα. Ε, έτσι είναι τα πράγματα. Κάτι το οποίο βέβαια δεν γίνεται κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε πως θα πρέπει να υπάρχει και κάποια δυνατότητα εφαρμογής, ίσως με, κάποια, με κάποιον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Και δεν το συζητήσαμε και αυτό και νομίζω έχουμε μια διαδικασία εδώ και ε, δύο-τρία χρόνια Αλλά τι συμβαίνει χάρη, για πράγματα οποία έχουμε ήδη εφαρμόσει και ισχύουν υποτίθεται για τις μικρές ε, υποθέσεις, εμπρότους αγώ στην ε, κάτω Σαξονία, δεν έχει γίνει τίποτα μετά από δύο χρόνια. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το συζητήσουμε τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η νομική ασφάλεια είναι μια ωραία λέξη, αλλά τι σημαίνει. νομική ασφάλεια σημαίνει αστικός κώδικας. Αυτό πάνε να πει νομική ασφάλεια. Αν ρυθμίσουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι, πάλι ένα κομμάτι έχουμε ρυθμίσει. Δεν είναι νομική ασφάλεια αυτό. Έχουμε μερική νομική ασφάλεια. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Οπότε θα πρέπει να περιοριστούμε σε μερικά βασικά θεμελιώδη πράγματα για να ξέρουμε τι είναι μια σύμβαση, πότε έχει συναυθεί μια σύμβαση, τι συμβαίνει κτλ. Και πολύ παραπέρα δεν θα πάμε. Γιατί, όπως σας είπα, το θέμα είναι μετά η εφαρμογή η οποία δεν θα πάει πολύ παραπέρα. Δικαίως θεωρούν τα κράτη-μέλη, εμείς όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε, όπως σας είπα, μέχρι τις 31 ε, Ιανουαρίου εξακολουθεί να υπάρχει η διαβούλευση της Κομισιόν, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να λάβουμε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων, ίσως με μια αξιολόγηση αντικτύπου ε, των πολλών, πολλών ε, ενδιαφερομένων, νομίζω. Οπωσδήποτε θέλουμε να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα προστασία των καταναλωτών. Μιλάμε γενικά για εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς οπωσδήποτε είμαστε αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα. Οπότε δικαίως ασχοληθήκαμε μαζί με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αλλά ρυθμίζουμε τόσα πολλά ε, ζητήματα από καταναλωτική πίστη μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, ασχοληθούμε και με κάποια βασικά ζητήματα να τα ρυθμίσουμε πραγματικά. Ας περιοριστούμε στο ενοχικό δίκαιο. Ξεκινήσουμε από εκεί. Σε... Στο 4-3-1, δηλαδή να κάνουμε μια στενή ερμηνεία, να μην πάμε πολύ μακριά, γιατί η εμπειρία μου μου λέει πως δεν θα ε, περάσουμε κάτι τέτοιο. Οπότε ας σκεφτούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε στην πράξη ως αρχές και να μην ε, θελήσουμε να ασχοληθούμε ολόκληρο το ενοχικό δίκαιο και τις ε, εξοδικαστικές στους εξοδικαστικούς συμβασμούς κτλ. Δεν γίνονται όλα αυτά, δεν θα λειτουργήσουν. Πρέπει να δουν πράγματα τα οποία έχουν όντως αποδεχτεί στην πράξη. Ευχαριστώ. Uh, uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσω το χρονοδιάγραμμα που έχω μπροστά μου, που βεβαίως ε, εξαρτάται από την συμφωνία με την... Ε, με την ε, αρμόδια επιτροπή. Ε, λοιπόν, 21 Ιανουαρίου θα το εξετάσουμε, υποβολή τροπολογιών 1η Μαρτίου το μεσημέρι και 22 Μαρτίου θα το εξετάσουμε στην Επιτροπή. Έτσι θα έχουμε τις ε, τροπολογίες μας ε, για την Νομική Επιτροπή τον Απρίλιο ώστε να ενσωματωθούν εκεί στην ε, έκθεση και να ψηφιστεί η έκθεση στην Ολομέλεια τον Μάιο. Συμφωνείτε? Είναι νέο, νέο χρονοδιάγραμμα. Το προηγούμενο ήταν πολύ πιο σφιχτό και, λίγο μπουρδα. Να τα πούμε έτσι απλά. Τόσο καλύτερο είναι αυτό, αλλά στο δούμε λίγο με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Γιατί εμείς έχουμε και ακρόαση, πράσινη βίβλο. Οπότε, εάν είναι η διαβούλευση να επηρεάσει τίποτα, δηλαδή αυτά τα οποία θεωρούν οι πολίτες μας, στους οποίους υποτίθεται εκπροσωπούμε, ας περιμένουμε και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Οπότε, πούμε, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Ε, well, I mean, I, I'm rather agree with you, but of course... Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά βέβαια το χρονοδιάγραμμα το ορίζει η νομική επιτροπή και όχι εμείς. Εσείς είστε υπεύθυνο για το ντοσιέ, θα περιμένουμε να μας ενημερώσετε. Να σας ευχαριστήσω όλους. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Να σα θυμίσω ότι η επόμενη μα συνεδρίαση θα είναι σε δύο εβδομάδες, στι 25, 3η 25 και 4η 26 Ιανουαρίου. Και όπως ήδη γνωρίζετε, την Τετάρτη 26 το απόγευμα έχουμε μια ψηφοφορία για την οδηγία για τη δικαίωμα του καταναλωτή. Επίσης την Τρίτη 25 έχουμε στρογγυλή τράπεζα για πιο αποτελεσματική και δίκαιη ε, αγορά λιανικής έκθεση για την οποία είναι η η κυρία Κοράτσα Μπέλτ και το πρόγραμμα δεν είναι πλήρες. Θα μπει στο site μας συντόμως και να θυμίσω και ίσως και να θυμίσω και στους θεατές μας που ίσως μας παρακολουθούν στο ίντερνετ ότι αυτή είναι η τελευταία εκδοχή αυτής της καταπληκτικής έκδοσης ε, του newsletter της IMCO με ένα σύντομο μήνυμα δικό μου. Όσοι δεν έχετε υπογράψει για να γίνετε φίλοι του δικτύου της ΣΥΜΚΟ, καταρχήν μπορείτε να το κατεβάσετε από το website, και, αλλά μπορείτε και να το υπογράψετε ώστε να το λαμβάνετε τακτικά στο, στη θηρίδα σας, ώστε να ενημερώνεστε για όλες τις εργασίες της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε την απόψινή συνεδρίαση και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες.